Możemy ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι. Αντικαθιστώ τον κύριο Ντεκάστρο. Εγώ θα είμαι πρόεδρο σήμερα. Να επαναλάβω. Σας καλωσορίζω, λέει ξανά ο Πρόεδρος αντικαθιστώ τον κύριο Δεκάστρο σαν πρόεδρο, τον κύριο Πάολο Δεκάστρο. Έχουμε κάνει κάποιες αλλαγές στην ημερήσια διάταξη, να σας τις εξηγήσω. Να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη με τις κάτωθι αλλαγές, θα ήθελα. Σχόλια. Έχω κάποια σχόλια. Μεταδίδεται η συνεδρίασή μας διαδικτυακά. Και όπως είπα δεν μπορεί να παρίσταται ο κύριος Δεκάστρο και μου ζήτησε να τον αντικαταστήσω στην ε, Προεδρία. Αυτό ήταν το πρώτο που είχα να σας πω. Και ο κύριος Σιλβέστρη δεν θα μπορέσει να παραστεί. Το σημείο λοιπόν 3 της ημερήσιας διάταξης αναβάλλεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Το σημείο 3 λοιπόν αναβάλλεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Αποφασίσαμε δε να διεξαχθεί αύριο το απόγευμα τριμερής ε, διάλογος. Οπότε το σημείο 11, η γνωμοδότηση του κυρίου Ράμες για τους ελέγχους θα αναβληθεί μέχρι αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί λοιπόν θα συζητήσουμε τη γνωμοδότηση του κυρίου, της κυρίας Ράιμερς. Μετά έχουμε τον κύριο Ρόντερς, το θέμα για την επιστημιστική κρίση και σημείο 13 την κατάσταση με τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής και αυτά έχουν αναβληθεί. ταυτόχρονα να σας πω ότι έχουμε διερμηνία σε όλες τις γλώσσες της Επιτροπής μας. Λοιπόν, ας πάμε στο σημείο 4 της σημερινής διάταξης. Προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών. Ο κ. Φαϊμών είναι ο εισηγητής. Θα γίνει μια ανταλλαγή απόψεων. Η πρόταση εδράζεται από το άρθρο 43 και έχει σκοπό να προστατεύσει την Ευρωπαϊκή Γεωργία και Δασοκομεία αποφεύγοντας την είσοδο και διάδοση ε, ξένων παρασίτων. και θέλουμε να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των διαφόρων φορέων και είναι κάτι που συνδέεται με την πρόταση για την παραγωγή αναπαραγωγικού υλικού και τη διάθεσή του στις αγορές. Είναι κάτι που αφορά τη γεωργία ε, ευρέως, την παραγωγικότητα του γεωργικού τομέα, τη δυνατότητα να διατίθενται προϊόντα στους καταναλωτές και να εξασφαλίζεται και ένα έσοδο για τους ε, αγρότες. Ε, είναι σημαντικότατο και δυσκολότατο ζήτημα. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τον εισηγητή, τον κύριο Φαϊμόν, να κάνει μια εισαγωγή στο δύσκολο αυτό θέμα. Σας δίνω λοιπόν το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας παρουσιάσω το σχέδιο κανονισμού για τα προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την αναθεώρηση νομοθεσίας στον τομέα και σήμερα έχουμε την πρώτη δυνατότητα να συζητήσουμε το σχέδιο κειμένου. Η έκθεσή μου θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και μετά θα διατεθεί σε όλους σας ούτως ώστε να υποβάλλετε τροπολογίες. Η προθεσμία για την υποβολή των ε, τροπολογιών είναι η 6η Δεκεμβρίου του 2013 και μετά θα ψηφίσουμε την έκθεση. Στόχος της νομοθεσίας είναι να αυξηθεί η προστασία κατά των επιβλαβών οργανισμών που πλήττουν τα φυτά σχε... Ε, σχετίστηκε με την οδηγία για τους σπόρους και το αναπαραγωγικό υλικό των φυτών ε, αποφασίσαμε αυτοί οι οργανισμοί να μπουν σε άλλο κανονισμό, τα επιβλαβείς οργανισμοί, ούτω ώστε να βελτιώσουμε την ευελιξία στον τομέα τη ε, της καταπολέμησης αυτών των επιβλαβών οργανισμών. Η νομοθεσία θέλει να, να ε, καλύψει το πρόβλημα αυτό. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να λαμβάνει προληπτικά μέτρα στον τομέα αυτό, ούτω ώστε να μπορεί να προστατεύονται έναντι τρίτων χωρών για μια τετραετία. Αυτή η χρονική περίοδος είναι απαραίτητη για να γίνει μια αξιολόγηση των κινδύνων. Το σχέδιο κανονισμού αναφέρει ότι οι πιβάτες που εισάγουν ελεγχόμενα φυτά στις αποσκευές τους απαγορευμένα φυτά, ή μάλλον αυτά πρέπει να υποστούν έλεγχο, θα πρέπει να συμμορφώνονται οι επιβάτε με του περιορισμού και του κανόνε τη αγωγή των φυτών. Το σχέδιο κανονισμού υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να διεξάγουν ελέγχους για τυχόν ύπαρξη παρασίτων σε περιοχές που δεν είχαν και αν εντοπιστούν σε κράτη-μέλη τέτοιοι επιβλαβείς οργανισμοί θα πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την εξάλληψή τους τα κράτη-μέλη. Μετά θα υπάρχει και υποχρέωση να διενεργούνται έλεγχοι και μέτρα εξουδετέρωσης αν αυτό χρειαστεί. Ε, και θα υπάρχει και προτεραιότητα όσον αφορά τους επιβλαβείς οργανισμούς. Θα έχει τη δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλλει ε, απομόνωση, καραντίνα, ε, κατά οργανισμών που δεν μπορούν να εξαλειφθούν. Και οι επαγγελματίες του τομέα θα πρέπει να καταχωρούνται σε ένα επίσημο μητρό και για την μετακίνηση φυτών υποχρεωτικά θα πρέπει να εκδίδονται φυτογειονομικά διαβατήρια που θα αποδεικνύουν ότι υπάρχει πλήρη συμμόρφωση με την νομοθεσία. Αυτά τα φυτογειονομικά διαβατήρια θα απαιτούνται για όλα τα φυτά για φύτευση και ε, θα εξηγείται ποια φυτά θα πρέπει να καλύπτονται από την έκδοση αυτού του διαβατηρίου. Όμως θα υπάρχει εξαίρεση για μικρές ποσότητες φυτών που θα απολούνται άμεσα στους τελικούς χρήστες. Δεν είναι σαφές όμως το πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να εναρμονίσει αυτή την εξαίρεση. Ε, Πλουστευμένο, τυποποιημένο φυτογειονομικό διαβατήριο θα πρέπει να εκδίδεται από συγκεκριμένου φορείς προκαθορισμένους. Η νομοθεσία συμπεριλαμβάνει κανόνες για τους παραγωγούς ξύλινων συσκευασιών. Αυτοί οι έμποροι θα πρέπει να επεξεργάζονται τη συσκευασία την ξύλινη και θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα διεθν... το Διεθνή Φυτογενομικό Κανόνι παριθμό 15 και να το αποδεικνύουν. Αυτό το σχέδιο κανονισμού θα οδηγήσει σε μεγαλύτερο διοικητικό άχθος για τα κράτη-μέλη και τις επιχειρήσεις και σε κάποιες περιπτώσεις τα θετικά αποτελέσματα είναι αμεληταία. Παραδείγματο χάρη, η υποχρέωση να αποστέλλονται αιτήσιες εκθέσεις όσον αφορά συμβάντα για καραντίνα, άρθρο 17 ή άρθρο 18 ή άρθρο 20 παράγραφος 3. Επίσης, εκθέσεις όσον αφορά τα αποτέλεσμα προσωμιώσεων ε, θα πρέπει να καταρτίζονται για οργανισμούς που έχουν προτεραιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 25.3. Θα πρέπει να συντάσσονται και εκθέσεις όσον αφορά τις πληροφορίες για επιβάτες, για πελάτες, ταχυδρομικές υπηρεσίες και όλα αυτά σε σχέση με την απαγόρευση εισαγωγής. Άρθρο 43, παράγραφος 3. Αυτές λοιπόν οι υποχρεώσεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και είτε να απλουστευτούν είτε να διαγραφούν. Διαβλέπω ένα πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει περισσότερες εξουσίες όταν θα υιοθετεί κατά εξουσιοδότηση πράξης και θα καθορίζει την συχνότητα διεξαγωγής προσωμιώσεων, κάτι που αναφέρεται στο άρθρο 25 ή όσον αφορά την ευαισθητοποίηση, οι εξουσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους τομείς αυτούς θα πρέπει να επανεξεταστεί. Πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να επανεξετάσουμε τη δυνατότητα οι επιθεωρητές να μπορούν να μπαίνουν σε ιδιόκτητα οικόπεδα και κτήματα για να εξαφανίσουν αυτούς τους επιβλαβείς οργανισμούς. Υπάρχει η δυνατότητα να επιτρέπεται σε επαγγελματίες όχι μόνο να εκδίδουν διαβατήρια για τα φυτά, αλλά να πρέπει να αποδεικνύουν την καλή υγεία των φυτών που διαθέτουν στην αγορά. Αυτό δυνάμει το άρθρο 82. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξηγήσει υπό ποιε προποθέσει οι εμπορευόμενοι που έχουν άδεια να διενεργούν αυτά τα επαγγελματικά καθήκοντα, πώς θα επιλέγονται. Το όλο εγχείρημα έχει στόχο την εξέβρεση πόρων. Χρειάζονται χρήματα αν θέλουμε να είναι πιο αυστηροί οι ισχύοντες κανόνες και να είναι πιο υψηλή προστασία κατά των ε, παρασίτων των φυτών. Για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να διαθέσουμε τους κατάλληλους πόρους. Το ίδιο ισχύει για τη χρηματοδότηση στον τομέα της υγείας των ζώων. Πιστεύουμε επίσης ότι θα πρέπει να χορηγείται μια οικονομική αποζημίωση για τους επαγγελματίες σε δικαιολογημένες ε, περιπτώσεις. Ε, μας αναφέρεται ότι συμπεριλαμβάνεται στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο αυτή η χρηματοδότηση οι προπτικές, τις προπτικές για το 2020 μέχρι το 2020 μάλλον. Αυτά έχω να πω στο περιπλοκότατο αυτό ζήτημα και προσβλέπω στην συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο, Και τώρα μπορούμε να αρχίσουμε τη συζήτηση με έναν γύρο ερωτήσεων. Κύριο Σάγκνιο, θέλει πρώτο το λόγο. Πρόεδρε, διαδικαστικό. Νομίζω ότι προηγείται η κυρία εδώ στα αριστερά μου. Θα θέλατε να λάβετε εσείς πρώτο το λόγο. Α, όχι. Μας είπατε για αυτές τις ασθένειε των φυτών και συμφωνώ ότι ο συνάδελφος που έκανε την εισαγωγή, την εισήγηση του τα βλέπει λίγο διαφορετικά από μένα, αλλά να σας πω ότι καταρχήν, εάν έχουμε τόσο υπέροχο θεσμικό όργανο όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι πάνε όπου θέλουν και όλα είναι τέλεια, τότε πάρα πολύ εύκολα να το δουν οι ασθένειε. Όμως, θα ήθελα να το δούμε από κάποια διαφορετική οπτική γωνία. Είναι πολύ επίκαιρο αυτό. Δεν προστατεύει τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση τα, τα, τα, τα φυτά. Ο ιδιωτικός τομέας και οι επιστήμονες το κάνουν που έχουν τα κατάλληλα φυτοφάρμακα που έλεγχουν την κατάσταση και πρόκειται για τεράστιες επενδύσεις οπότε αυτοί θα έπρεπε να δικαιούνται να προσδοκούν κάποιο είδους ε, αξιόπιστο και υπεύθυνο νομικό πλαίσιο από τους πολιτικούς αφέντες οπότε θα πρέπει όλα αυτά να έχουν θεμέλιο την επιστήμη και όχι την πίεση από τα λόμπι ούτε την ε, μόδα. Τους τελευταίους μήνες είδαμε τους επιστήμονες να χάνουν το δάσο τα πόδια τους διότι εμείς συμφωνήσαμε ότι αυτό το φάρμακο που σκοτώνει τις μέλισσες πρέπει να απαγορευτεί το είπαν, το είπαν οι επιστήμονες και είπαν τελικά οι ότι αυτό θα γίνει από του χρόνου και αυτό θα έχει πάρα πολλές φορές συνέπειες. Εγώ, ξέρετε, είμαι γεωργός. Και έχω τέσσερα εκτάρια που τα φύτεψα να Ανθίσαν τον Αύγουστο και ήταν, μπορείτε να φανταστείτε πόσες, πόσες μέλισσες ήταν γεμάτο αυτό το χώρο. Δηλαδή, επόμενα μπορεί να δείτε ότι πριν γίνει η απαγόρευση αυτού του φυτοφάρμακου που τη σκοτώνει έχουν ήδη ανακάμψει. Σήκωσαν κεφάλι με τους. Οπότε βλέπετε ότι δεν είναι λογικό να, να, να βιαζόμαστε να απαγορεύσουμε προϊόντα. Μόλις τώρα, λέει ο πρόεδρος, μου είπαν ότι έχουμε ένα σωρό Μέλισσα, ότι είναι μια χαρά η ή οπότε βλέπουμε τον Επιτρόπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής, ο οποίο θα μα μιλήσει πάνω σε αυτό. Αλλά πρώτα πρώτα δώσουμε το λόγο στην κυρία Αγίουσο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει που τη σειρά που να πάρουμε τον λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί μα είπε τόσο λεπτομερό όσον αφορά το σχέδιο κανονισμού. Αυτό είναι κομμάτι από αυτή τη δέσμη μέτρων. Είναι πέντε κανονισμοί και πρόκειται να αντικατασταθούν έτσι 700 νομοθετικές πράξεις σε σχέση με τον έλεγχο, με τις εισαγωγέ που έχουν να κάνουν με, τη, με τα φυτογειονομικά και με τα κτηνιατρικά. Ε, έχει καταβάλει προσπάθεια η Κομισιόν, αλλά το πράγμα είναι πολύ δύσκολο. Δύσκολο κανείς να είναι πολύ αποτελεσματικό. Όλα αυτά είναι πολύ πολύ περίπλοκα. Σας λέω αυτές εξ αρχής ότι σε αυτή την πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγράφει πάρα πολύ τις εκτελεστικές πράξεις και τις ε, κατεξιοδότηση πράξεις. Τα λέει πάρα πολύ ξεκάθαρα και συγκεκριμένα ο βασικός κανονισμός. Δεν χρειάζεται κανείς να προσφύγει σε τέτοια νομοθετήματα σαν τις κατουσιοδότηση πράξης. Λέμε λοιπόν εδώ πέρα Ποιο έχει τι αρμοδιότητα, την επαγρύπνηση κλπ. Τα φυτογενομικά. Άρα, επί τη βάση του προσυγχρονισμού, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ορίσει ποιε θα είναι οι αρμόδιε αρχέ οι οποίε θα πρέπει να ασκήσουν αυτή την υποπτία, αυτόν τον έλεγχο. Είναι ξεκάθαρο αυτό, αλλά θα πρέπει να εξαθαρίσει και η Κομισιόν του βασικού κανόνε του παιχνιδιού. Και να ζητηθεί από τα κράτη-μέλη να υποδείξουν τις αρμόδιες αρχές για επαγρύπνηση και έλεγχο. Έτσι θα είμαστε πιο πρακτικοί και πιο αποτελεσματικοί. Άλλο. Τι είναι με αυτούς τους ε, φόρους για τις μικρές επιχειρήσεις, τους μικροσυναλλασσόμενους, αυτό σηκώνει συζήτηση, αλλά όχι στα πλαίσια αυτού του κανονισμού. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να φορτώσουμε στους ευρωπαίους παραγωγούς με περισσότερα. Ήδη έχουν πολλά βάρη οικονομικά να φέρουν. Κάτι άλλο το οποίο αφορά πολύ την Ισπανία. Εξαιρεί η Επιτροπή τα κανάλια τον κανονισμό και θεωρεί ότι πρέπει να έχουν μεταχείριση τρίτης χώρας. Είναι αλήθεια ότι στην ισχύουσα οδηγία ε, προβλέπεται κάτι για τα Κανάρια. Αλλά είπαμε ότι σε έξι μήνες μετά από τον κατάλογο των ε, ασθενειών τότε θα γίνει προσαρμογή γιατί τα Κανάρια όπως όλα τα νησιά βρίσκονται σε μια ιδιαίτερη κατάσταση. Θα πρέπει μόνος κανείς να είναι πολύ προσεκτικός. Έχουν βέβαια τα Κανάρια ε, για την πιστοποίηση, για τις αρρώστιες, έχουν τη, τη δική τους νομοθεσία. Αλλά μάλλον θα πρέπει εδώ πέρα να καλυφθούν από αυτό το νομοθέτημα. Να μην έχει τη μεταχείριση τρίτης χώρας γιατί αυτό εμποδίζει την πρόσβαση των προϊόντων των Καναρίων στην ευρωπαϊκή αγορά. Θέλω να νομοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις ε, εισαγωγές. Νομίζω ότι εδώ το θέμα είναι ευρύτερο. Η Ένωση θα πρέπει να προστατευτεί γιατί έχουμε ενιαία αγορά, οπότε τα προϊόντα και το αναπαραγωγικό υλικό κυκλοφορούν ελεύθερα απ' και μπουν σε μια χώρα. Αλλά αυτό το οποίο εξάγει κάθε χώρα σε τρίτε χώρε, αυτό είναι θέμα εθνικό. Θέμα διμερών συμφωνιών. Φέτο, α πούμε, έχουμε 200 πρότυπα διαφορετικών πιστοποιητικών. Τρίτων χωρών που έχουν επίδραση επί ημών. Ο κάθε χώρα θα πρέπει να προστατεύεται για το τι εισάγεται στην Ένωση. Βασικά αυτά ήθελα να σας πω. Ωραία, λοιπόν περιμένουμε το κείμενο της έκθεσης και μετά, ως συνήθως, θα υποβάλουμε προπολογίες. Και τώρα δώσουμε το λόγο στην κυρία Ράιμερς. Διαβάζοντας αυτή την έκθεση και βλέποντας και το συνολικό πακέτο, είδα, γιατί μιλάμε για πολλές εκθέσεις, είδα ότι ε, προβλέπονται πάρα πολλά είδη. Νομίζω ότι ακούμε πολλά παραπονά στην πράξη για το πώς θα γίνει αυτό, πώς θα οργανωθεί όλη αυτή η δουλειά και πραγματικά πρέπει να σκεφτούμε πόσες είναι αυτές οι διατάξεις που ζητούνται από την Κομισιόν. Θέλει η Κομισιόν να ρυθμίσει τα πάντα. Η πρακτική όμως και οι συνήθειες της ε, χώρες μέλη της Ένωσης δεν λαμβάνονται υπόψη και νομίζω ότι ε, δεν υπάρχουν συστήματα κινήτρων. Μιλούμε για ασθένειες, μιλούμε για επιβλαβείς οργανισμούς, για τα φυτά. Ε, Υπάρχουν κάποιες ασθένειες όμως που η ε, πρώτη που, ε, που του συμβαίνει δεν, ε, δεν θέλουν καν να το δηλώσουν ότι έχει υπάρξει κάποια ασθένεια στα δικά τους φυτά γιατί θεωρούν ότι δεν θα υπάρξει κάποια αντιστάθμιση. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει και ένα κίνητρο. Αυτοί που πλήττονται πρώτοι να μην αρχίζουν απλώς ε, να ε, κρύβουν ή να καίνε τα φυτά τους αυτά επειδή φοβούνται ότι θα ε, υπάρξει τεράστια οδηγητικό άφθος μέχρι να καταλήξουν σε κάποιο αντιστάθμισμα. Θα πρέπει να, να τους δοθούν κίνητρα έτσι ώστε εγκαίρως να μπορούν να δράσουν, ειδικά όταν ανακαλύπτουν την ασθένεια των φυτών. Νομίζω ότι είναι καλό που λέμε τουλάχιστον ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πιο σύγχρονε τεχνικέ. Και αντί να μιλούμε για βουνά χαρτούρας που πρέπει να μεταφέρονται, να, πηγαίνει, να πάμε σιγά σιγά σε πιο ηλεκτρονικέ πηγές, να μπορούμε να σκανάρουμε, να υπάρχουν κάποιοι κωδικοί, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η δουλειά. Και επίσης, όσο πιο πολύ θέλουμε να ελέγξουμε τόσο πιο πολύ προσωπικό θα χρειάζεται κανεί στη διοίκηση για να ελέγχει, χρειάζεται, χρειάζεται προσωπικό στι εταιρείε για να εκδώσουν τα πιστοποιητικά, τα διαβατήρια κτλ. Οπότε πρέπει να δούμε και το θέμα τη αναλογικότητα σε σχέση με αυτά που ζητούμε. Πρέπει να, είμαστε, να έχουμε μια ισορροπία. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και χαίρομαι που την κάνουμε, γιατί σίγουρα θα υπάρξουν πολλέ καλέ προτάσει. Κάτι άλλο να σημειώσω. Μιλούμε για την υγεία των φυτών. Δεν μιλάμε για προστασία ζώων ή για προστασία φυτών. Χαίρομαι που χρησιμοποιούμε την, θέματα όπως ε, η κλωνοποίηση, η γενετική, η τεχνική κτλ. για να τα συζητήσουμε, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το πακέτο, πάρα πολύ ιδιαίτερο, πάρα πολύ τεχνικό. Μίλησε και ο συνάδελφος πριν για, τον, για την νέο νοικοτινοίδη δεν ε, νομίζω ότι θα καταφέρουμε να το ολοκληρώσουμε ένα τόσο εξειδικευμένο και περίπλοκο θέμα να το ολοκληρώσουμε. Είμαστε σε πίεση χρόνου ούτως ή άλλως, οπότε καλό θα ήταν να λειτουργήσουμε ε, σωστά και με αν θέλουμε βεβαίως να το κάνουμε αυτό. Και επίσης να πω ότι μιλούμε για διάφορες ε, κατηγορίες φυτών, οι οποίες δεν μπορούν πάντα να θεωρούνται ίδιες σε ό,τι αφορά και την αποθήκευση και τη μεταφορά τους κτλ. Δεν μπορούν λοιπόν οι κανόνες να είναι ομοίοι για όλα τα είδη φυτών. Θα πρέπει να έχουμε ξεχωριστούς. Ευχαριστώ. Το Πολύ πρακτική η προσέγγιση σας και βλέπω ότι εμβαθύνουμε περισσότερο σε αυτόν τον πολύ περίπλοκο τομέα. Νομίζω ότι θα συζητήσουμε περισσότερο και στα πλαίσια της ακρόασης για το θέμα αυτό. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Μποβέ. Euh, θα ήθελα να προσπαθήσω να είμαι συγκεκριμένος. Δυστυχώς έχουμε δραματικά παραδείγματα στην Ευρώπη περιπτώσεων που δεν βρήκαν λύση και καταστράφηκαν εκατοντάδες ε, χιλιάδες τρέματα όπως μια ασθένεια που είχε το όνομα Σάρκα, Σάρκα και έπληξε τα δέντρα στην Νότια Γαλλία. Δεν εισήχθη από πολιτές φυτών, αλλά από τη δημόσια έρευνα, την επιστημονική έρευνα. Ποτέ δεν ρύθμισε το πρόβλημα η Ευρωπαϊκή Ένωση και αποζημίωση των γεωργών ε, έγινε μεγάλες δυσκολίες. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα με αυτή την ασθένεια στη Γαλλία Υπάρχει σχετισμός με τη Ρουμανία και ανησυχώ πολύ για τη Ρουμανία με αυτή την ασθένεια που την πλήττει επίσης. Είναι σημαντικά θέματα. Δεν αφορά μόνο τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και η δημόσια έρευνα θα πρέπει να σέβεται τους κανόνες του παιχνιδιού. Άλλο είδος ασθένειας που ίσως απειλήσει τις νήσους Καναρίους πολύ σύντομα, αφορά τα απορροκευτικά, κατέστρεψε όλη την παραγωγή στη Φλόριδα και βρίσκεται και στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή. Το πρόβλημα αυτών των ασθενειών είναι ότι δεν υπάρχει ε, λύση εκτός από την εκρίζωση. Και είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να λαμβάνετε υπόψη, που είναι καινούριο. Η αύξηση θερμοκρασίας, η αλλαγή του κλίματος. Αυτή η αύξηση οδήγησε σε μετακινήσεις αυτών των προβλημάτων και έχουμε πραγματικό πρόβλημα. Οι ασθένειες αυτές δεν είναι μόνο πρόβλημα που δημιουργείται από το εμπόριο, αλλά με την αλλαγή των τόπων παραγωγής. Πρέπει να δούμε πώς γίνεται η παραγωγή σε σχετισμό λοιπόν με τις ασθένειες αυτές. Τέλος, να πω ότι στους τρόπους παραγωγής υπάρχουν πραγματικοί κίνδυνοι. Σήμερα στις χώρες χρησιμοποιούν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και υπάρχουν αντιστάσεις κάποιων εντόμων. Και έχουν γίνει πάρα πολύ ανθεκτικά τα έντομα λόγω των γενετικά τοποποιημένων οργανισμών. Έχουμε και τέτοιου είδους προβλήματα, δεν είναι ασθένειες που δημιουργούνται και εμφανίζονται από συγκεκριμένο πρόβλημα συνδέονται με τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Που κάνουν, δημιουργούν αυτά τα υπερέντομα, τα πολύ ανθεκτικά έντομα που δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τα παραδοσιακά μέσα. Ε, και αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη σαν ζητήματα εντός της όλης της λογικής ανάλυσης. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Δεν είναι ζητήσει άλλη το λόγο. Επομένως, να μας πει τώρα εκπρόσωπος της Επιτροπής ή εκπρόσωπος, η κυρία Σιμεών. Μπορείτε να απαντήσετε κυρία τις ερωτήσεις. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Επιτροπής σας για τα όσα είπαν. Όσον αφορά την πρώτη παρατήρηση, αφορούσε περισσότερο την προστασία των φυτών και των συναφών προϊόντων και αυτό τόνισε και η κυρία Ράιμαρ. Όμως αυτά τα προϊόντα, τα σχετικά με την προστασία των φυτών, δεν υπάρχουν σε αυτό το νομοθέτημα. Υπάρχονται σε ένα διαφορετικό πλαίσιο νομικό και κανονιστικό. Εδώ, προκειμένου δεν θέλουμε να ασχοληθούμε με κάποιου τέτοιε αγωγέ, θεραπείε. Τώρα, όσον αφορά τι εφαρμοστικέ, εκτελεστικέ και κατεξουδότηση πράξη που ήταν αντικείμενο άλλη παρατήρηση, είπατε ότι αυτό απαιτέρεσε κατάχρηση σε αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό το οποίο έχουμε εδώ, έχουν, θέλουμε να έχουμε ένα βασικό νομοθέτημα το οποίο να θέτει κάποιε αρχέ. Και αυτέ οι αρχέ να ενσωματώνται στο βασικό νομοθέτημα και στα παραρτήματα. Και παραπέρα να έχουμε τις τεχνικές λεπτομέρειες οι οποίες να περιέχονται σε κατοξιοδότηση ή σε εκτελεστική πράξη. Βέβαια, κατά την κατάρτιση αυτών των κατεξοδότηση πράξεων είχαμε διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες και τις εκτελεστικές πράξεις θα έχουμε την επιτροπολογία που θα μας βοηθήσει. Θα μπορέσουμε να λάβουμε τα πιο δόκιμα μέτρα. Οπότε και σας διαβεβαιώ ότι δεν πρόκειται να κάνουμε του κεφαλιού μας. θα βασιστούμε σε ό,τι λένε οι εμπειρογνώμονες, σε ό,τι προκύψει από την επιτροπολογία. Τώρα όσον αφορά τι θα καλύψει αυτός ο κανονισμός, θέλουμε να καλύψουμε κάποιες γεωγραφικές περιοχές. σε σχέση με την προέλευση κάποιων ε, ασθενειών. Εξαιρούμε ότι δεν ανοίξει αυτή την ε, περιοχή που θέλουμε να καλύψουμε. Ε, αυτές οι περιοχές που ξέρουμε έχουν άλλα είδη, άλλα είδη φυτών κλπ. Και έτσι θα φροντίσουμε καλύτερα την κυρίω επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά έτσι, δημιουργείται η πιθανότητα σε εκείνες τις περιοχές να προστατευθούν από κάποιες ασθένειες που ενδημούν στην επικράτεια της Ένωσης. Concerning the economic incentive to, to report outbreaks of pests for... Όσον αφορά το ξέσπασμα αυτών των ασθενειών, κάποιος το είπε προηγουμένως. προβλέπονται αντισταθμίσεις, αποζημιώσει για διάφορου από του συναλλασσόμενου όσον αφορά την καταστροφή του φυτικού κεφαλαίου. Είπαμε ότι αυτό είναι βασικό κίνητρο για εκείνου για να αναφέρουν σχετικώ και να λαμβάνουν τα μέτρα που χρειάζονται αρκετά νωρίς για την καταπολέμηση των ασθενειών Και υπάρχει το κανονιστικό πλαίσιο και για τα κτηνιατρικά και για τα φυτογενομικά κλπ. Και για τα ε, φυτοαναπαραγωγικά. I think that uh, these are the main uh, comments that uh, I wanted. Αυτά είναι τα βασικά που είχα να σας πω προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να σας πω ότι θα διεξαχθεί ακρόαση στις 26 Νοεμβρίου. Τροπολογίες μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου και τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου κανονικά πρέπει να γίνει η ψηφοφορία. Επίσης, θα γίνει και ανάλυση της ε, γνωμοδοτήσεως. Εάν δεν υπάρχουν σχόλια, θα γίνει ανάλυση λοιπόν της εκθέσεως. Θα ήθελα να πάμε στο σημείο 5 λοιπόν. Φυτικές επιλογές. Ποιες είναι οι επιλογές για την αύξηση της ποιότητας και της παραγωγής. Θα γίνει μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά την έκθεση. Είναι έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας και αφορά την αναπαραγωγή των φυτών, όπως προανέφερα, αφορά τις επιλογές για την αύξηση της ποιότητας και της παραγωγής. Αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας ανατέθηκε στην κυρία Πάουλσεν. Θα ήθελα να της δώσω το λόγο, να... έχει το λόγο Μαρίτ και κάνε μας μια παρουσίαση του θέματος. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρέπει να πω ότι σχεδόν λυπάμαι που είναι στην ημερήσια διάταξη σήμερα το θέμα αυτό, διότι δεν αποτελεί ένα κομμάτι του πακέτου ε, για τους ελέγχους που παρουσιάστηκε πριν. Απλώς εδώ ε, εκφράζω τη δική μου ιδέα που συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση πρωτοβουλίας Βλέπετε, συνεργάζομαι πολύ στενά με το Βασιλικό Ινστιτούτο Γεωπονίας στη Στοκχόλμη και συνέχεια εκεί τίθεται διάφορα ζητήματα ε, για την έρευνα, για την ανάπτυξη, για τη δημιουργία ποικιλιών φυτικών και γίνεται ένα θέμα που αφορά και τις διατλαντικές σχέσεις και γίνεται ζήτημα που αφορά και τις πολυεθνικές που ελέγχουν την αγορά. Θα ήθελα να πω ότι ανέλαβα αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας διότι θεωρώ ότι η Ευρώπη πρέπει να ανακτήσει τον έλεγχο της ανάπτυξής της στον τομέα. Όλοι μας σε αυτή την Επιτροπή γνωρίζουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Γεωργία και θα αντιμετωπίσει τα επόμενα 30-40 χρόνια. Με την αύξηση του πληθυσμού πρέπει να αυξήσουμε την παραγωγή τροφίμων. Κατά 70% περίπου. Ξέρουμε ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται με λιγότερη ενέργεια, λιγότερη γη, λιγότερα νερά, ε, λιγότερα χημικά κλπ. Όλα αυτά βέβαια ε, δημιουργούν πιέσεις και απαιτήσει ε, για, τη δημιουργία διαφόρων ποικιλιών φυτών. Πρέπει να βρούμε τρόπο για την αύξηση της σοδιάς στην ίδια αρρώσιμη γη που διαθετούμε. Πρέπει να βρούμε σοδιές, φυτά που να αντέχουν να αντέχουν είτε περισσότερο νερό, είτε περισσότερη ξηρασία, υψηλότερες θερμοκρασίες, νέα παράσιτα, νέες ασθένειες κλπ. Άρα οι προκλήση είναι τεράστια. Θα ήθελα λοιπόν αυτό να το συζητήσουμε. Δεν ξέρω αν όλοι έχουμε εδώ κάποια λύση έτοιμη, αλλά θα πρέπει να γίνει προσπάθεια και έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειάζεται ένας συντονισμός των προσπαθειών όσον αφορά την έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα που διατίθεται για την έρευνα, για αυτό το σκοπό. Θέλουμε και υποστήριξη της ποικιλομορφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα. Οι μικρές επιχειρήσεις όλο και περισσότερο χάνουν έδαφος διότι οι κανόνες, οι διατάξεις και τα χρήματα όλα πηγαίνουν στις μεγάλες, πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και τις πολύ μεγάλες εκμεταλλεύσεις. Και επηρεάζονται εξελίξεις από τη δική τους επιθυμία να αλλάξουν ε, αυτά που καλλιεργούν, τα φυτά που καλλιεργούν και γιατί θέλουν να προωθήσουν τα χημικά που διαθέτουν. Θέλω να επιστρέψουμε σε μια ευρωπαϊκή βιοπικιλότητα, να χρησιμοποιήσουμε την ε, σύγχρονη τεχνολογία για αυτόν τον σκοπό. Ανέλαβα λοιπόν αυτή την πρωτοβουλία, διότι θεώρησα ότι τελειώνουν διαπραγματεύσεις για την επόμενη επταετία της κοινή αγροτικής πολιτικής, άρα θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε το επόμενο στάδιο. Ποιες είναι οι εξελίξεις που θέλουμε, που θέλουμε να πάμε. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας, τι έχετε να πείτε εσείς για όλα αυτά. Αυτό δεν σχετίζεται πλέον με την πρώτη ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι αποκλειστικά μια έκθεση ίδια πρωτοβουλία. Αυτά είχα να σα πω. Ωραία, να ξεκινήσουμε τώρα τη συζήτηση. Η κυρία Λεμπρούν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα από πλευρά τη πολιτική μα ομάδα να χαιρετήσω την πρωτοβουλία τη ε, Άννα Μαρία Πόλσεν σε σχέση με την επιλογή αυτή, τη φυτική. Πάρα πολύ βασικό θέμα. Και διαπιστώνουμε πάντες πώς η, ζήτηση πρόκειται με το 2050 να αυξηθεί κατά 70% όσον αφορά ε, αυτού του είδου τα, τα, και λοιπά, τι ανάγκε των φυτών. Είναι θέμα παγκοσμίας δημογραφίας κατά κάποιο τρόπο και βλέπουμε ότι αυτό αφορά την άνοδο του επίπεδου, αλλά βέβαια υπάρχει και θέμα ζήτηση ε, του κρέατος που συνδέεται με αυτό. Και έχουμε χρειάζονται 15 κιλά σιτηρών για να παράξουμε ένα κιλό κρέας. Οπότε τα πράγματα είναι απλά. Θα πρέπει να παράξουμε περισσότερο. Εάν θέλουμε να είμαστε πρωτοπόροι στα αγροδιατροφικά. Και αν επομένω δούμε τι προοπτικές υπάρχουν, τότε διαπιστώνουμε ότι τα αγροδιατροφικά είναι το κλειδί για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την οικονομία, για γενικά για την διαστατική ισορροπία. Επομένως το να βράξουμε περισσότερα δεν σημαίνει βέβαια να παράξουμε ό,τι να είναι. Θα γράψουμε την λοιπόν, υπόψη τι πόρους έχουμε, θα πρέπει να συμφιλιώσουμε την παραγωγικότητα με την βιωσιμότητα, την αηφορία. Αυτό απαιτεί ο κόσμος. Οπότε υπάρχουν σημαντικέ προσπάθειες που καταβάλλονται όσον αφορά τον τομέα του περιβάλλοντος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δείξει ότι αυτέ οι προοπτικέ οικονομικά και κοινωνικά είναι βιώσιμε. Πάντως ε, σήμερα όλοι η προβληματική συμπυκνώνεται στο ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να επιστρέψουμε ό,τι έχουμε από πλευρά ε, έρευνα για να μπορέσουμε να έχουμε λύσεις νέε, εναλλακτικέ, να τα αποκρίνονται τις ανάγκε τη κοινωνία, αλλά και τη αεφορονάπτυξη. Άρα αυτό θα πρέπει να γίνει. Η εφορία με την παραγωγικότητα να μην είναι αντίθετε για άλλη μια φορά να αποδείξουμε ότι συμβαδίζουν. Από τη μια μεριά να παράγει κανεί περισσότερο, από την άλλη μεριά να παράγει καλύτερα. Τύπος παραγωγής, τύπος καλλιέργεια, οπότε φτάνουμε στην, στο θέμα αυτό στις φυτικές επιλογέ. Πρόκειται για ένα θέμα τεράστιο. Αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα το πλαισιώσουμε χωρίς να βγούμε εκτός θέματος όπως είπε ο Ζωζέ Μποβέ κάπως τα λέει διαφορετισμένα, θα πρέπει να τα λέει πιο συγκεκριμένα αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα χρησιμοποιηθούν κάποιες χημικές ουσίες να χρησιμοποιήσουν όσο γίνεται καλύτερα τις φυσικές ε, διεργασίες και θα πρέπει βέβαια να δοθούν κίνητρα στους Ευρωπαίους ούτως ώστε να μπορέσουμε να προστατευτούμε τον διεθνή ανταγωνισμό. Για να έχουμε γεωργία ποιοτική θα πρέπει να της δώσουμε τα μέτρα, τα μέσα προστασίας και έτσι να αναδειχθεί η γεωργία μας. Δεν θα ήταν φυσιολογικό ούτε καλό να, περιθωριοποιηθούμε στο θέμα αυτό ξέρω τι είναι με τα μεταλλαγμένα κλπ. Τη βιοτεχνολογία. Ξέρουμε ποιες είναι οι απόψεις των Γεωργών. Θα πρέπει να ακούσουμε τις απόψεις όλων, όλων των μπλεκομένων κλάδων. Και έτσι να με προσοχή, να επαγρυπνούμε. Γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας ως βουλευτών να διρεμήσουμε το ζήτημα μέσω γίνεται περισσότερη δίκαιη κρίση. Καινοτομία, πολύ σημαντική, από πάντοτε. Επομένως, θα πρέπει πάντοτε να αμφισβητούμε αυτά τα οποία έχουμε δεδομένα και να διερευνούμε κάθε φορά την γενετική πολυμορφία. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσουμε να λύσουμε αυτό το θέμα πια δεν παίρνει αναβολή. Ευχαριστώ. πολύ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στην Μποβέ. Νομίζω ότι η δουλειά που κάνει η κυρία Απόλσεν, ακόμα και αν πρόκειται για νομοδότηση την ώρα, θα προωθήσει θα ταράξει κάπως την Επιτροπή, να βγει από τη βεβαιότητα στην οποία βρίσκεται. Ο προπολογισμό στην έρευνα είναι το συγκεκριμένο μπορούμε να εντοπίσουμε. Τα τελευταία χρόνια είχαμε προπολογισμό ή την έρευνα που είχε σαν στόχο αποκλειστικά τις επιχειρήσεις για να γίνουν αποδεκτοί οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί από τον πληθυσμό. Θα θυμούνται κάποιοι ένα πρόγραμμα trans Food 12 εκατομμύρια ευρώ για να καταπιούν και να χωνέψουν τους, τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς οι Ευρωπαίοι. Δεν δούλεψε και τα 12 εκατομμύρια ευρώ μπήκαν στη τσέπη των επιχειρήσεων. Τι προτείνω λοιπόν στην έκθεση να προτείνουμε μέσω του προπολογισμού για την έρευνα σε σχέση μεταξύ Επιτροπής Γεωργίας και Επιτροπής Έρευνας να καταρτιστεί χρηματοδότηση για τη συμμετοχική έρευνα για την παραγωγή σπόρων, συνεργασία δηλαδή μεταξύ παραγωγών και ερευνητών. Ξεκινώντας από, την, από τα χωράφια και τα, να δούμε ποια εδάφη υπάρχουν, πώς επιλέγουν τους σπόρους οι γεωργοί ανάλογα με το χώμα, να συνεργαστούν με τους ερευνητές για να αναπτυχθούν ε, συμμετοχικοί τρόποι ανταλλαγής των σπόρων να βγούμε από την νέα παραγωγή σπόρων που ισχύουν για όλα τα εδάφη χωρίς την παραμικρή προσαρμογή στο έδαφος. Το πραγματικό πρόβλημα που έχουμε σήμερα και το λέω αυτό απαντώντας ανησυχία της κυρίας Λεμπρέν είναι ότι σήμερα οι σπόροι είναι όλοι ισοδύναμοι ανεξάρτητα από το χώμα, ανεξάρτητα από το κλίμα, όλοι οι ίδιοι είναι. Βάζει κανείς την κατάλληλη ποσότητα νερού και τα χημικά. Διαφορετικά δεν υπάρχει σοδιά. Θα πρέπει να αντιστρέψουν τη διαδικασία. Ξεκινάμε από το έδαφος, από το κλίμα, από την πραγματικότητα και θα παράγουμε τους πόρους που αντιστοιχούν σε αυτές τις ανάγκες. Είναι μια καινοτομία αυτή. Όσον αφορά την αντίληψη της έρευνας. Δεν στρέφεται κατά της έρευνας. Ξεκινά από το υπάρχον δυναμικό και όχι αντίστροφα. Τυποποιημένη προσέγγιση. Πολύ δουλειά πρέπει να γίνει. Αν γίνει θα προχωρήσουμε. Πρέπει να εξετάσουμε την νομοθεσία που συζητείτε. Δεν τελείωσαν συζητήσεις, αλλά θα δημιουργήσει πρόβλημα αυτή η νομοθεσία. Η νομοθεσία για τη σπορά, για τους σπόρους. Που επιτρέπει επιχειρήσεις πάντα να διατηρούν τον έλεγχο και δεν επιτρέπει στους γεωργούς να ανταλλάσσουν τους σπόρους τους. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Αρνιού. Άγνιου. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Το ερώτημα της κυρίας Πόλσον ήταν πολύ απλό. Ποιε είναι οι δυνατότητε που έχουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα των εσοδιών. Έχουμε αρκετέ. Καταρχά, μπορούμε να διασταυρώσουμε τι ποικιλίε, έτσι ώστε να, είναι βρούμε, να έχουμε κάτι καλύτερο από, από τους Δεύτερον, η, διασταύρωση των φυτών. Έχουμε την ποικιλία Α και την ποικιλία Β και θεωρούμε ότι υπάρχει κάποιο αδύναμο κρίκο στον Α, αλλά η ποικιλία Β το έχει, αλλά μπορεί να το αντιμετωπίσει και αν συνδυάσουμε τις δύο αυτές ε, ποικιλίε μπορούμε να έχουμε ένα, ένα μια καλύτερη ποικιλία. Βέβαια μπορεί κανείς να, λάβει, να έχει και πολύ χειρότερα αποτελέσματα, δεν το ξέρουμε. Ε, μια άλλη επιλογή είναι να βάλουμε σπόρους μέσα σε ένα σακούλι και να κρεμάσουμε αυτό το σακούλι και να κάψουμε αυτούς τους ε, σπόρους και μετά να θεωρήσουμε ότι θα υπάρξει κάποια, ε, κάποιος εκφυλισμός ε, ο οποίος θα μεταλλάξει αυτούς τους σπόρους. Ε, μετά, κάπως έτσι βέβαια ε, έφτιαχνε φαγητό και ο Φραγκενστάιν. Αλλά αυτό εντάξει δεν μας ανησυχεί. Αυτό που ανησυχεί όμως όντως είναι ότι οι επιστήμονες μπόρεσαν να απομονώσουν ένα γονίδιο σε κάποιο φυτό κάποιες ποικιλία και μπορούν να το ε, μεταφέρουν πολύ συγκεκριμένα ε, σε κάποιο άλλο φυτό. Βέβαια, το πράσινο λόμπι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι αυτό είναι πάρα πολύ κακό ε, και ότι όλοι θα είμαστε σκλάβοι στους κακούς καπιταλιστές. Δεν τα έχετε ακούσει αυτά. Αποκλείεται. Έχουμε πολύ καλούς επιστήμονες στα βρετανικά εργαστήρια και ένα από αυτά στο Ρόθενστετ, στο Hertfordshire, ε, οι επιστήμονες λοιπόν εκεί ε, βλέπουν τα πράγματα πάλι από την αρχή για το πώς μπορούμε με νέους τρόπους να ελέγξουμε τα έντομα. Ε, αντί να, σκοτώσουμε τα έντομα που έρχονται στα φυτά, ενισχύουν την, την ανοχή τους. Ε, αποτρέπουν τα ε, έντομα ε, να πάνε να, να πλήξουν κάποια φυτά. Έγιναν λοιπόν κάποιες προσπάθειες να να αντιστραφούν τα αποτελέσματα μια δίκη που έγινε πέρσι τον Μάιο. Ε, ήρθαν αρκετοί μάρτυρε, Εγώ πήγα υπέρ τη ε, για την υπεράσπιση των Βρετανικών εργαστηρίων. Αυτοί οι 150 άνθρωποι που ήρθαν θεώρησαν ότι δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την αστυνομία και όλου εμά που πήγαν να υπερασπιστούν την ιδέα αυτή. Γι' αυτό αποφάσισαν ότι θα πρέπει να, κάνουν, να βγάλουν κάποιου πύριου ε, αντικαπιταλιστικού λόγου και ξεκίνησαν να το κάνουν. Αυτή λοιπόν είναι η στάση. Ε, δεν νομίζω ότι η Ευρώπη έχει δικαιοδοσία να ε, ε ελέγξει εδώ. Γίνεται, καθίστανται όλα πολύ πιο, ε, πολύ πιο περίπλοκα, πολύ πιο ακριβά και θα πρέπει να επιτρέψουμε αυτό τον τομέα πολιτική να εξελιχθεί από μόνο του. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν από μόνα του πώ θέλουν να χρησιμοποιήσουν την γενετικώ τροποποιημένη τεχνολογία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα πολύ ενδιαφέροντα τα πολύ ενδιαφέροντα σας σχόλια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Πόλσεν που υπέβαλε αυτή την έκθεση. Είναι περίπλοκη και σημαντική. Να πω ότι ποια είναι η θέση του κυρίου Καπούλα Σάντο, που είναι σκιώδη ηγητή. Μου ζήτησε ω εκπρόσωπο τη ομάδα των Σοσιαλιστών να εκφράσει την άποψή του γενικές τοποθετήσει, γιατί είναι η αρχή τη συζήτηση, βέβαια. Λέει ότι η βελτίωση φυτική συμπεριλαμβάνει διάφορες τεχνικές που έχουν σαν στόχο να επηρεάσουν τη διαδικασία ανάπτυξης των φυτών, ούτω ώστε να αναπτυχθούν ποικιλίε ανώτερες ανάλογα με τη θεσιμότητα. Με ανώτερες ποικιλίε εννοούμε ποικιλίε με, με ανώτερη απόδοση ή που αντιστάνται καλύτερα στις διάφορες εξωτερικές συνθήκες, κλίμα, έδαφος κλπ. Αυτή η βελτίωση παράγεται ανεξάρτητα από την πρακτική τη σχεδιασμένη και είναι συνέπεια της πρακτικής των παραγωγών φυτών που κάνουν φυσική, προκαλούν μια φυσική επιλογή. Από την άλλη πλευρά έχουμε την επιλογή που κάνει η βελτιωση παραγεται ανεξαρτητα απο την πρακτικη τη σχεδιασμενη και ειναι συνεπεια της πρακτικης των παραγωγων φυτων που κανουμε φυσικη προκαλούμε φυσικη επιλογη απο την αλλη πλευρα εχουμε την επιλογη που κανει η βιοτεχνολογια ο τρόπος με τον οποίο γίνεται επιλογή όμως επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της φυτικής ποικιλία μακροπρόθεσμα. Βιωσιμότητα σε επίπεδο, όπως και η παγκοσμιοποίηση, είναι λέξη της μόδας και χρησιμοποιούνται καταχρηστικά. Και χάνουν την έννοιά τους αυτές οι λέξεις. Θα ήθελα λοιπόν να προσπαθήσω, λέει ο συγητής, να δούμε τι εννοούμε βιωσιμότητα όσον αφορά τη φυτική ποικιλία. Πρέπει να συνδυάζει αυτή η ανταγωνιστική παραγωγή χωρίς απώλεια γενετικής ποικιλία μακροπρόθεσμα. Μπορεί να είναι ελκυστικό αυτό εμπορικά για τους γεωργούς, δηλαδή στις καλλιέργειές τους να καλλιεργούν περισσότερο με ποικιλία. Μακροπρόθεσμα όμως αυτό θα έχει συνέπειες ε, που δεν αντιστρέφονται όσον αφορά τη διαθέσιμη βιολογική ποικιλία. Και είναι αντιστόφως ανάλογη αυτή η βιοποικιλότητα με τον κίνδυνο της απερίμωσης των καλλιεργιών. Διότι αν υπάρχει μονοκαλλιέργεια γίνονται πολύ ευάλωτε. Εμείς που παίρνουμε τις αποφάσεις πρέπει να δημιουργήσουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο. Ούτω ώστε η φοιτική επιλογή να γίνεται σε αυτό το πλαίσιο. Να λάβουμε υπόψη υπεύθυνη ρεαλιστική προσέγγιση που ανταποκρίνεται τι σημερινέ ανάγκε χωρί να υπονομεύει τι επόμενε γενιέ. Πρέπει να επαγρυπνούμε. Να δεχτούμε τι επιστημονικέ εξελίξει Χωρί να λησμονούμε όμω τι συνέπειε που έχουν οι επιλογές μας μακροπρόθεσμα. Γνωρίζουμε ότι θέλουμε σταθεροποίηση τη απόδοση τη παραγωγή και γίνεται λόγω τη αλλαγή του κλίματο πιο ευάλωτη η παραγωγή. Και από παράλληλα ζητούμε και μεγαλύτερη παραγωγή τροφίμων. Μην λησμονούμε ότι η πρόσφατη κρίση των τιμών οδήγησε σε ελλείψει σε κάποια μέρη του κόσμου μόνο. Η φυτική επιλογή, συμβατική ή μέσω μοριακής προσέγγισης μπορεί να δώσει απαντήσεις. Θέλουμε ληστική προσέγγιση όμως. μονούμε τη μικροβιολογία των εδαφών και άλλες μεταβλητές. Να λάβουμε υπόψη και την αρχή της πρόληψης. Χωρίς να τη χειραγωγούμε, υπεύθυνα να τη λάβουμε υπόψη. Να βρούμε τη σωστή ισορροπία στις λύσεις που θέλουμε να βρούμε και απαιτούνται. Δεν θέλουμε να υπονομεύσουμε όμως τη δυνατότητα παραγωγής για τις μελλοντικέ γενιές. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να υποστηρίξω την έκθεση της κυρίας Πόλσεν. Είναι πολύ πατριωτικό από μέρους της να ερευνά αυτό το θέμα. Όλες οι αποχρώσεις που ανέφεραν και οι συνάδελφοι είναι απολύτως ε, συμβατές με το θέμα αυτό και θα ήθελα να ε, συμφωνήσω με αυτό που είπε ο κ. Μποβέ. Εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πολύ διαφορετικές χώρες με πολύ διαφορετικές συνθήκες και πολύ συχνά μια εταιρεία που έχει ζητήσει να γίνει μια έρευνα έχει κάνει δοκιμές, έχει δει ότι θα μπορέσει να υπάρξει κάποιο οικονομικό κέρδος, έχει ξεκινήσει την διαφήμιση εντός και της Ένωσης. Ε, ταυτόχρονα όμως, αυτό το προϊόν μπορεί να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλα κλίματα. Και έτσι οι γεωργοί πιστεύουν ε, αυτή τη διαφήμιση, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες ε, εκμεταλλεύσεις, αγοράζουν το προϊόν, το χρησιμοποιούν, δεν βγαίνει τίποτα και κανένα δεν τους ε, αποζημιώνει για το κόστος και για τα έξοδα που έκαναν. Πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε στο ότι τα, η καλλιέργεια των φυτών και η δημιουργία νέων ειδών θα πρέπει να ε, τροποποιηθεί και να προσαρμοστεί στι ε, περιφερειακέ συνθήκε. Και κάθε χώρα μπορεί να το κάνει αυτό, για να, γιατί η ίδια η χώρα ξέρει ποιε είναι οι συνθήκε τη για να προωθήσει ναι, την ναι. καλλιέργεια. Ε, στην, ε, στην ε, Λετωνία πρόσφατα ε, μια, μια εταιρεία η οποία ασχολείται με την καλλιέργεια πατάτας και με ενημέρωσαν ότι υπάρχουν διάφορα είδη πατάτας τα οποία έχουν καλλιεργηθεί στην Λετωνία και είναι πολύ καλά, ναι. είναι πολύ ανθεκτικά σε, διάφορα, ε, σε διάφορους επιβλαβείς οργανισμούς, δίνουν καλές οδιές και έχουν χρησιμοποιηθεί, έχουν χρησιμοποιηθεί για πολλά χρόνια στην Λετωνία. Και μετά βλέπω ότι τέτοια είδη, τέτοιο είδο πατάτας χάνουν πολύ σύντομα τα καλά του στοιχεία. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τι πρακτικές δοκιμές που γίνονται πάνω σε αυτά τα είδη. Και επίση πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μιλούμε για την ισορροπία μεταξύ της ελεύθερης αγοράς και της ποιότητας των τροφίμων. Θυμούμε πριν από ε, πολλά χρόνια όταν ε, ε, αυτοί, οι πατάτες που έτρωγα εγώ τότε δεν συγκρίνονται με αυτές που τρώμε σήμερα, ούτε σε ποιότητα ούτε σε γεύση. Τώρα είναι σκληρέ, δεν έχουν καμία γεύση, δεν έχουν το άρωμα της πατάτας. Δεν λέω ότι πρέπει να πάμε πίσω στο παρελθόν, αλλά θα πρέπει να δούμε το θέμα της ποιότητας θα πρέπει ίσως να ξεχωρίσουμε ποιες είναι οι εταιρείες που ασχολούνται με βιολογικούς τρόπους παραγωγής. Θα πρέπει να δούμε και το θέμα της συσκευασία ίσως. Αυτά τα προϊόντα μπορεί βεβαίως να είναι πιο ακριβά. Γιατί ε, οι φτηνές ε, πατάτες ή φτηνές ντομάτες που δεν σου δίνουν την απαραίτητη, δεν έχουν την απαιτούμενη θρεπτική αξία, δεν είναι καλά ποιοτικά προϊόντα. Ελπίζω λοιπόν να έχουμε αποτελέσματα μέσω και αυτής της έκθεσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι, είναι αλήθεια ότι δεν ήμασταν μικροί οι ε, εύσεις ήταν διαφορετικές, αλλά μήπως τα νιάτα ήταν η αιτία. Τέλος πάντων, να δώσουμε τώρα το λόγο στην εκπρόσωπο, στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Γιάννη Καμιστήσο. Τον κύριο Καραμίτσο. Thank you, uh, uh, Mr. Chair. Κυρία Καραμίτσο, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, θα σας μιλήσω αντί του κυρίου Καραμίτσου. Mm. Ο κύριος Καραμίτσος είναι ο αρμόδιος γιατί είναι τεχνικό το θέμα που αφορά την αναπαραγωγή των φυτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τις προκλήσεις αυτές που δημιουργούνται από την ε, αλλαγή του κλίματος και από το, το αυξανόμενο πληθυσμό των φυτών φυτά και ακριβώς ε, τον, τον πληθυσμό της γης και τα, ε, τα διατροφικά ζητήματα σε σχέση με το πόσο Σημαντικό είναι να καταπολεμηθούν τα προβλήματα που προκύπτουν. Άρα θα πρέπει να διατηθούν χρήματα για έρευνα προς αυτό το μέτωπο. Είναι καινοτόμος αυτός ο κλάδος με την αναπαραγωγή ε, των φυτών από τους πιο καινοτόμους μάλιστα. Επίση. έχουμε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών μία έρευνα σχετικά. Μα ληφθεί αυτό υπόψη κυρίως να βρει μικρότερες καλλιέργειες. Ίσως τώρα δεν φωτίστηκε αρκετά η πραγματική εικόνα για το πώς έχει η κατάσταση για την αγροτική στην Ευρώπη σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Έχουμε πάρα πολλές ε, εκμεταλλεύσεις μικρές και μεγάλες. Και ιδίως όσον αφορά τα φρούτα, ακόμη περισσότερο. Εμείς τώρα έχουμε μια μελέτη τόσο ώστε να ξεκαθαριστεί το τοπίο. Δεν έχουμε μόνο μεγάλες εταιρείε. Έχουμε μικρομεσαίες. Και θεωρούμε ότι η σημερινή νομοθεσία όσον αφορά τη θέση εμπορία των σπόρων πραγματικά θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις αυτές. Έτσι θα υπάρχουν δικαιότητες για συνταγωνισμό. Το Σεπτέμβριο θα έχουμε να δούμε προς τα μπρος έχουμε λοιπόν, αυτή την πρόταση για τι ποικιλίε που θα πρέπει να καταχωρηθούν σε κάποιο μητρό πριν τεθούν σε εμπορία. Προτείναμε μια καινούργια διαδικασία, τόσο να υπάρχει ε, για τις δοκιμές, μια νέα διαδικασία. Use of new So this testing is out in members. Οπότε να με τον καιρό, το κλίμα που κρατεί σε κάθε χώρα, ρυθμίζεται η καλλιέργεια να παραγωγή του φυτού. Η αντίσταση, η ανθεκτικότητα στις ασθένειες, οι ανάγκες σε φυτοφάρμακα, ανάλογα με το αν θα πρέπει να έχουμε λοιπόν, πιο ανθεκτικά φυτά ή όχι σε διάφορα φαινόμενα ή σε ασθένειες. Έχουμε το υλικό τώρα, το προπλησιαστικό που θα ρυθμιστεί και έχουμε προτείνει διάφορες προσεγγίσεις καινούργιε. Στην πρόστασή μας προσπαθούμε αυτούς που ασχολούνται και με τους κήπους και με τις υπόλοιπες καλλιέργειες να τους πλαισιώσουν. Αυτή η δοκιμή των ποικιλιών στα κρατημέλια έχει επίσημο χαρακτήρα. Τα κρατημέλια έχουν αυτούς τους, τους καταλόγους των ε, συστάσεων και έτσι οι καλλιεργητές έχουν ε, αμερόληπτες ε, αντικειμενική πληροφόρηση για τη χρήση των ποικιλιών. ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν δεν υπάρχουν σχόλια, θα ξαναδώσω το λόγο στην εισηγήτρια αν θα έχει την καλοσύνη να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις που ετέθησαν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Πόλσον. Πρέπει να πω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένη διότι ακούσαμε πολλές και ποικίλε απόψεις. Αυτό είναι κάτι πολύ δημιουργικό. Στις 5 Νοεμβρίου θα γίνει μία ακρόαση. Θα συμμετάσχουν τρεις ερευνητές. Ένας θα αναφερθεί στις τεχνικές αναπαραγωγής που υπάρχουν σήμερα. Ίσως ήταν καλό να τις γνωρίζουμε. Και να μπορούμε να αποφασίσουμε υπέρ ή κατά. Θα έχουμε και Αμερικανό ερευνητή βιοτεχνολόγο που όμως ασχολείται με βιολογικές καλλιέργειες, καλός συνδυασμός. Πολύ καλή αρχή θα είναι αυτή. Και θα πρέπει να συνεχίσουμε τη δημιουργική μας αυτή προσέγγιση. Είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της συζήτησής μας. Και τα συμπεράσματα θα ακολουθήσουν πολύ αργότερα μετά τις συζήτησεις μας. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια, λέει ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι η ακρόαση αυτή θα είναι χρησιμότατη για τις εργασίες μας. Στις 25 Νοεμβρίου θα γίνει ανταλλαγή απόψεων. Έχουν προθεσμία για τις τροπολογίες 2 Δεκεμβρίου και αυτό το θέμα μπορεί να ψηφιστεί από την Επιτροπή Ιανουάριο ή Φεβρουάριο ίσως. Ορίστε. Ζητώ συγγνώμη. Λέει κυρία Πόλσον, θέλω να πω ότι ήδη βλέπετε το άλλο θέμα, την ακρόση για την υγεία των ζώων. Μάλλον μπερδευτήκατε κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρος. Ναι, θα συζητήσουμε τώρα το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Που είσαστε ξανά η μας για αυτό το θέμα, κυρία Πόλσον, αφορά την υγεία των ζώων είναι η τρίτη αναθεώρηση του νομοθετικού πακέτου για τα φυτογενομικά και την υγεία των ζώων. Το, αυτό το τμήμα αφορά την υγεία των ζώων. Το ευρωπαϊκό κεκτημένο αποτελείται από 50 κανονισμούς και οδηγίες και περίπου 400 νομοθετήματα δευτερογενούς νομοθεσίας. Κάποια νομοθετήματα έχουν υιοθετηθεί από το 1964. η νομοθεσία για την υγεία των ζώων θέμα το οποίο θα συζητήσουμε θέλει, έχει σκοπό να έχουμε προστευμένη ενιαία διαφανή σαφή προσέγγιση, σαφές πλαίσιο για την υγεία των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγγήτριά μας είναι η αντιπρόεδρος μας η Μάριτ Πόλσον. Μάριτ, έχει το λόγο. Είναι η μέρα στο σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα συζητήσουμε το ένα κομμάτι του πακέτου ΣΑΝΚΟ. Σε αυτή τη θητεία θα πρέπει να τοποθετηθούμε επί του θέματος. Και από ό,τι φαίνεται θα μπορέσουμε έτσι να αντικαταστήσουμε 40 εφιστάμενες οδηγίες και κανονισμούς με το νέο πλαίσιο. Είναι περιπλοκότατο το έγγραφο νομικά. Το πρώτο που έχω να πω και να κάνω είναι το εξής. Θα ήθελα να πω ότι ανεξάρτητα από το πώς αντιλαμβάνεστε τον όρο υγεία των ζώων, δεν μιλάμε για νομοθεσία που αφορά τη συνολική υγεία των ζώων, αλλά είναι μια νομοθεσία η οποία αφορά μόνο τις ασθένειες, τις μεταδοτικές που πλήττουν τα ζώα. Μεταδοτικές ασθένειες αφορά η νομοθεσία όταν μιλάμε υγεία των ζώων. Δεν έχει καμία σχέση με τις ασθένειες των ζώων που δεν είναι άμεσα μεταδοτικές. Είναι δύσκολο να το έχει αυτό κανείς υπόψη του πάντα. Θα ήθελα λοιπόν να πούμε ότι εδώ μιλάμε για προστασία κατά των μετα... δηλαδή υγεία των ζώων, νομοθεσία για την υγεία των ζώων και αποφυγή διάδοσης μεταδοτικών ασθενειών. Όταν μιλάμε για την υγεία των ζώων, αναφερόμαστε σε πολλούς φορείς. Και πώς μάλλον θα αντιληφθούν οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι φορείς, θα θεωρήσουν ότι μιλάμε για την ε, καλή ζωή, για την ε, ε, καλή υγεία των ζώων εν γέννη. Δεν πρόκειται γι' αυτό. Τέλος πάντων, σε επιστρέψω τώρα στο τι κάνει ακριβώς η νομοθεσία. Η, ανα... οδηγία αφορά τις διάφορες καταστροφές. Δηλαδή, αν έχουμε αυτό πυρετό, πυρετό των χείρων, και λοιπά διάφορες ασθένειες. Όταν συζητούμε τις μεταδοτικές ασθένειες, 70% από αυτές είναι κοινέ και για τους ανθρώπους και τα ζώα. Και μόνο το 30% από αυτές τις ασθένειες αφορούν μόνο τα ζώα. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτές οι ασθένειες μπορούν να δημιουργήσουν πραγματικές καταστροφές για τους ανθρώπους, για τα ζώα, για τις κοινωνίες και την οικονομία. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε σαφέστατη σχετική νομοθεσία και ένα ξεκάθαρο σύστημα για τον εντοπισμό και για την πρόληψη των ασθενειών για να αποφύγουμε τη διάδοσή τους, τη μετάδοσή τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, πάντα το έχουμε υπόψη μας. Πάμε τώρα στις διάφορες περιπλοκές και τις αντιφάσεις που υπάρχουν. Όταν διαβάζει κανείς την προτινόμενη νομοθεσία, ανακαλύπτει ότι σχετίζεται με εφαρμοστικέ πράξεις και καταξιοδότηση πράξης. Συνεχώς. Σχεδόν κάθε παράγραφος αναφέρεται σε αυτές τις πράξεις. Ξεκινάει λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το δικαίωμα να λάβει την ανοσχετική απόφαση, να λάβει αποφάσεις για τα πάντα. Από τη μορφή των εγγράφων μέχρι τις ασθένειες που πρέπει να καταχωρούνται, ποια είδη ζώων πρέπει να συμπεριλαμβάνονται κλπ. Αυτό είναι πρόβλημα. Διότι είναι θέμα επιστημονικό, είναι θέμα γνώσεων. Είναι θέμα του να μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει νέες ασθένειες. Να μπορεί κανείς να αντιδρά γρήγορα. Δεν μπορούμε να έχουμε λοιπόν νομοθεσία η οποία εξαρτάται συνεχώς από κατεξουσοδότηση πράξης. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα περιθώριο για επιστημονική προσέγγιση, τεχνική προσέγγιση, γρήγορες αποφάσεις, χωρίς να χάνουμε τον έλεγχο εμείς. Αυτή είναι μία από τις επιπλοκές του ζητήματος. Η άλλη περιπλοκή, επιπλοκή μας, συγγνώμη, πρέπει να συζητήσουμε, είναι από τη μια θέλουμε την ελεύθερη εσωτερική αγορά και ελπίζουμε ότι με την οικονομική κρίση και με την ψηλή ενέργεια τη σημερινή ότι πραγματικά θα καταφέρουμε να αναπτύξουμε την εσωτερική αγορά. Αυτό από το ένα χέρι θέλουμε την ελεύθερη αγορά. Απ' την άλλη βέβαια το εμπόριο ζών των ζώων και το εμπόριο των ζωικών προϊόντων αυτό κάθε αυτό δημιουργεί κινδύνους μόλυνσης. Πώς θα χειριστούμε τη λειτουργία εσωτερικής αγοράς αποφεύγοντας όλες τις μεταδοτικές ασθένειες αυτή είναι η άλλη επιπλοκή που θα πρέπει να βρει λύση. Όσον αφορά την υγεία των ζώων και πώς να συμπεριφερόμαστε στα ζώα, αυτό αναφέρεται στην νομοθεσία που αφορά την βιολογική ασφάλεια. Έχει αυτό τον τίτλο, αφορά αυτό το θέμα. Βιοασφάλεια. Αυτό είναι σημαντικό διότι πρέπει να καταλάβουμε το εξή. Αν τα ζώα δεν τα προσέχουμε, αυξάνεται ο κίνδυνος ε, μόλυνσης. Αν μεταφέρονται υπό κακέ συνθήκες τα ζώα, τότε είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος μετάδοσης κάποιες ασθένειας. Πώς το κρίνουμε αυτό, πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό, πώς το χειριζόμαστε. Και άλλο ζήτημα που πρέπει να βρει λύση. Δεν βλέπω πώ όμω είναι το εξή θέμα. Τα αντιβιωτικά. Η αντίσταση που αναπτύσσεται κατά των αντιβιωτικών. Σε αυτή την νομοθεσία θεωρείται ως επικίνδυνη μεταδοτική ασθένεια. Και είναι πρόοδο το ότι συμπεριλαμβάνεται το πρόβλημα της αντίστασης αντιβιωτικά και θα προβληματιστούμε από αυτού. Αυτή η αντίσταση όμως στα αντιβιωτικά που οφείλεται στην κακή χρήση ή την κατάχρηση των αντιβιωτικών σχετίζεται με τις μη μεταδοτικές ασθένειες. Τα αντιβιωτικά χρησιμοποιούνται επί δεκαετίες. Σαν μια γενική αιγίδα κάλυψη ε, για να καλυφθούν προβλήματα στη διατροφή των ζώων, στην κτηνοτροφία. Να καλυφθούν τα προβλήματα της ελληπούς κτηνοτροφίας. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την αντίσταση στα αντιβιωτικά και την κατάχρηση των αντιβιωτικών όταν όλα αυτά τα κουβεντιάζουμε μόνο στο πλαίσιο των μεταδοτικών ασθενειών. Ανέφερα, πιστεύω, τις μεγαλύτερες αντιφάσεις που βρίσκει κανείς στην προτινόμενη νομοθεσία και διαβάζοντάς τη έχετε υπόψη ότι γενικά είναι ένα θέμα διαφόρων ελεγκτικών συστημάτων, διαφόρων τύπων ελεγκτικών συστημάτων. Ε, δεν είναι θέμα βιολογίας. Δεν είναι θέμα πρακτικής ε, χειραγώγησης, ε, προσέγγισης των ζώων. Είναι περίπλοκο νομοθετήματα, από τα δύσκολα νομοθετήματα, 257 παραγράφους συμπεριλαμβάνει. Ηράκλειο το έργο που μας περιμένει και φοβούμε ότι θα δεχτούμε χιλιάδες αντιπροτάσεις που δεν θα σχετίζονται με αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι της νομοθεσίας αλλά θα εντάσσονται στην ε, καλή μεταχείριση των ζώων εν γέννη και τη σχετική νομοθεσία. Διότι για μία ακόμη φορά αυτή η νομοθεσία συγκεκριμένη αφορά μόνο τις μεταδοτικές ασθένειες. Τίποτα άλλο. Είναι θέμα δημιουργία συστήματος ελέγχου που θα προλαμβάνει και θα χειρίζεται και θα αντιμετωπίζει και θα σταματά ε, Θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα. Ελπίζω ότι θα καταφέρετε να διαβάσετε όλη την πρόταση και ότι θα καταφέρετε ε, να είσαστε πλήρως ενήμεροι για τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Όντω είναι Ηράκλειο ο άνθρωπο μα. Να ευχαριστήσω την κυρία Συγκέντρια και να δώσουμε το λόγο στην κυρία Γκαρσία Πέρο θέλει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ επίση πάρα πολύ την κυρία Πόλσεν για την παρουσίασή τη. Έθεσε επιστραπέζει πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα για αυτή τη γενικότερη προβληματική σε σχέση με την καλομεταχείριση των ζώων και την υγεία τους γενικότερα. Τώρα, εκ μέρους της ε, συναδέλφου Μπαρατή που είναι η σκιώδης των σοσιαλιστές, να σας πω τι πρεσβεύει για το θέμα μας. Τις τελευταίες μέρες έχουμε λάβει τρεις ε, παρεμβάσεις από Ιταλία, Πορτογαλία και Αυστρία από τα Εθνικά Κοινοβούλια όσον αφορά αυτό το σχέδιο που έχει σχέση με την υγεία των ζώων. Ε, σε αυτές τις ε, παρεμβάσεις και προτάσεις να γνωρίζετε ότι η αρχή της επικουρικότητας έχει ε, τηρηθεί και υπάρχουν κάποιες εμβολίες να βρω ότι συνέχεια έχουμε εκτελεστικέ πράξεις και κατεξοδότηση πράξεις εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής οπότε συμφωνούν και αυτοί οι συνάδελφοι με τα όσα είπε η κυρία Πούλσεν. Επίσης εμείς σοσιαλιστές συμμεριζόμαστε αυτές τις αμφιβολίες οπότε έχει πάνω από 100 άρθρα αυτό το σχέδιο κανονισμού και δίνει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή ε, για τέτοιε ε, κατευθύντικέ πράξει και άλλα 50 άρθρα που τη δίνουν τη δυνατότητα για εκτελεστικέ πράξει και δεν λέει τίποτα όσον αφορά και τον κατάλογο των ασθενειών για τα οποία ισχύουν αυτά. Ε, όσον αφορά επομένω το βεληνικέ του οργανισμού, αυτό εμποδίζει. Οπότε αυτό είναι θέμα θεσμικό και πολιτικό που θα πρέπει να επιλύθει επίση το ότι έχουμε τόσε πολλέ κατηγορίε πράξει όσον αφορά στη δυνατότητα της Επιτροπής να, να πρέπει να απλουστεύσει την ισχύουσα νομοθεσία, θα πρέπει να γίνει πιο κατανοητή για τους ε, κτηνιάτρους, για τους ε, γεωργούς και για τους μεταφορείς των ζώων. Εν τέλει, αυτή η πρόταση, όπως είναι τυπωμένη σήμερα, δεν δίνει ένα πλαίσιο εις τον νομοθέτη για το πώς θα πολιτεύεται στο μέλλον. Γι' αυτό και η συγγετρία θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές σε αυτόν τον κανονισμό και έτσι ο κανονισμός να μπορέσει να έχει κάποια σημαντικά στοιχεία όπως ακριβώς ένα κατάλογο των ασθενειών ε, που ε, όπως έχει σήμερα κατάσταση είναι θέμα ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίσης ξέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έχει δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόσο ώστε υπό ορισμένες συνθήκες να μπορεί να παρέμβει με, με, με ιδιαίτερο και, και τρόπο, γιατί υπάρχουν πολλές φορές ιδιομορφίες, υπάρχουν ευαίσθητα λεπτά δύσκολα θέματα, όμως παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιες πτυχές του κανονισμού αυτού που θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο πολιτικής ρύθμισης και απόφασης του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου επίσης. Θα πρέπει να βρούμε ένα κριτήριο οργανωτικό όσον αφορά αυτές τις εξουσιοδότηση πράξεις και έτσι να δούμε πώς ε, αυτή η δυνατότητα αρμοδιότητα θα είναι ρυθμισμένη με τέτοιο τρόπο τόσο ώστε να είναι εύληπτη και απλή για όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται με τη γεωργία στην Ευρώπη. Επίσης θα πρέπει να είναι δυνατόν να δοθεί δυνατότητα στους ε, καταναλωτές στην Ευρώπη των τρίτων χωρών το πώς θα μπορέσουν να συμμορφώνονται όσον αφορά την παραγωγή κάποιων προϊόντων με αυτά τα οποία επιτάσσει η νομοθεσία μας φυτογενομικά κλπ. Ούτως ώστε να μπορούν αυτά τα προϊόντα να τεθούν σε εμπορία σε ξένες αγορές και έχω τώρα κατά νου συγκεκριμένα την αγορά των ΙΠΑ ε, διότι θα έχουμε συνομιλίες για την ε, Ένωση Ελευθερών Εμπορίου ΙΠΑ Ευρώπης. Κύριε η οποία στη Σαρτινή την περιφέρεια της ε, υποφέρει από την πανόλη των χείρων και άλλες αρρώστιες ούτως ώστε Αυτές μαστίζουν μόνο στην αγορά και τη δική μας και την Αμερικανική, οπότε νομίζουμε ότι τέτοιο κίνδυνο υπάρχει και για, και για άλλους ε, κτηνοτρόφους, αλλού στην Ευρώπη, οπότε αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. dziękuję pani poseł. tej zabierze głos pan poseł Ευχαριστούμε πολύ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Σμιτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ ήμουν ασκιώδη ε, και θα ήθελα να ευχαριστήσω, να συγχαρώ την κυρία Πόλσεν που πραγματικά είναι πολύ αποσχολημένη σήμερα. Είναι πολύ καλό που είναι αυτή η συγκέντρωση, σε αυτόν τον πολύ περίπλοκο φάκελο. Θα πρέπει να είμαστε πολύ πειθαρχημένοι λοιπόν στον τρόπο με τον οποίο θα τον αντιμετωπίσουμε και χαίρομαι που είπε και η Μαρίτα ότι ε, δεν μιλούμε για την ευζοία των ζώων εδώ, ε, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην βάλουμε διάφορα στοιχεία της ε, ευζοίας των ζώων σε τούτο τον φάκελο, γιατί δεν είναι αυτό το σημείο. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτός ο φάκελο έχει να κάνει κυρίως με την αντιμετώπιση και την απάλληψη των ασθενειών, των επιζωτιών. Ακούσαμε διάφορε ανησυχίε για τι καταξιότητε συμπράξει. Ε, η Κομισιόν νομίζω όμω ότι πήρε τη σωστή απόφαση ω προ αυτό αν θέλαμε πολύ πιο συγκεκριμένο πλαίσιο ευρωπαϊκό, ε, σημαίνει ότι δεν θα είχαμε ευελιξία για τα κρατημέλη και αυτό δεν θα ήταν εύκολο να εφαρμοστεί, θα κυρωνόταν από μόνο του. Ε, η διαφορά είναι ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει ε, αντίδραση από τα αρχέ των κρατών μελών, γιατί αυτέ είναι που θα εφαρμόσουν τα όσα πρέπει να γίνουν. Οπότε η συνεργασία του είναι απαραίτητη. Το έχουμε δει και σε άλλα θέματα, όπου καταραίουν τα πάντα επειδή οι αρμόδιε αρχέ δεν συνεργάζονται. Ακούσαμε κάποιε ανησυχίε, όπω είπα ήδη, από κάποια κράτη-μέλη, το μελετούν και τα κοινοβουλιά του η πρόταση όσα έχει δεν είναι η τελική. Νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να την βελτιώσουμε και να δούμε τι θα κάνουμε και με τις κατεξοδότητες συμπράξεις όταν θα προκύπτουν. Δύο πράγματα θα ήθελα εγώ να πω. Καταρχάς για τα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς. Νομίζω ότι είναι πολύ σωστή ιδέα, θα πρέπει να την δούμε, αλλά Ερώτημα για την Κομισιόν. Υπάρχει άλλη συζήτηση για το ποιος είναι ο προπολογισμό που έχουμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα εθνικά εργαστήρια να συνεχίσουν την εργασία τους και να μας δίνουν την εμπειρογνωμοσύνη που χρειαζόμαστε. Επίσης, είχα πει ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μην προσθέσουμε άχρηστες πληροφορίες σε αυτό το φάκελο. Ε, ας πούμε, τα, τα, ε, η σαλμονέλα, οι ασθένειε όπω οι, ζω, οι άλλε ζωονόσοι δεν αποτελούν τμήμα τούτη τη ε, έκθεση, ε, παρόλο που είναι μεταδόμενε ασθένειε. Νομίζω ότι η ευζοία των ζώων δεν ταιριάζει εδώ. Το να ε, μπουν όμω αυτά τα σημεία, τα αυτά τα τέσσερα για τι συγκεκριμένε ασθένειε. εδώ τούτο το φάκελο θα τον εμπλούτιζε θεωρώ. Προσβλέπω λοιπόν στην περαιτέρω δουλειά, είναι πολύ και την περιμένουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στην κυρία Γέμπλε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια, την κυρία Πόλσεν, για τα όσα έχει κάνει μέχρι τώρα και για τον πρώτο φάκελο. Συνεργάζεται πολύ στενά μαζί μας και την ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ και για την εισαγωγή σας, για τα σχόλιά σας. Ε, μας παρουσιάσατε πώς έχει το πακέτο, το περιγράψατε πάρα πολύ καλά. Αν θέλουμε τώρα να ακολουθήσουμε τον ε, δρόμο που μας ε, δείξατε και το έχετε συζητήσει με όλους τους κοιόδες, θεωρώ ότι στο τέλος θα έχουμε κάνει μια ωραία πρόταση ως κοινοβούλιο. Αυτά που αναφέρατε, τα σημεία που αναφέρατε και χαίρομαι που και οι υπόλοιποι σκιώδεις είναι της ίδιας άποψης. Τι θα κάνουμε δηλαδή με τις κατεξουδότητες πράξεις, με τις εφαρμοστικές πράξεις που υπάρχουν στην ε, πρόταση της Κομισιόν. Θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά ποιο αποφασίζει πότε και τι και με επιπίας βάσεως θα αποφασίζονται όλα αυτά. Και ένα δεύτερο σημείο σημαντικό επίσης είναι κάτι που θα πρέπει να είναι απολύτω σαφέ. Εδώ μιλούμε για προστατευτικά μέτρα για ασθένειε, μεταδιδόμενε ασθένειε. Μιλούμε δηλαδή για μια διαδικασία που θέλουμε να σταματήσει όταν μεταδίδονται οι ασθένειε. Και βεβαίω μιλούμε και για πρόληψη κρουσμάτων. Μιλούμε δηλαδή για πολλά στοιχεία τα οποία θα θέλαμε να συμπεριλαμβάνονται όντως θα πρέπει να ε, είμαστε προσεκτικοί, να μην προσθέσουμε πράγματα που δεν ανήκουν σε τούτο το φάκελο, αλλά που μπορούν να τύχουν καλύτερη ε, εξέταση σε άλλους φακέλους. Ας ε, μείνουμε εδώ στα σημαντικά. Θα ήθελα να πω επίσης ότι υπάρχουν κάποια σημεία που με ανησυχούν λίγο, τα άρθρα 5-8 για, για τον κατάλογο των επιζωτιών Μιλούμε για τις συνέπειες τη βιοπικιλότητα και την ε, ρήπανση του περιβάλλοντος. Αν μελετήσουμε αυτό το θέμα, δεν θα μπορούσαμε ίσως εδώ να... Δεν θα ανοίγαμε μια πόρτα ώστε να μπουν πράγματα εδώ που θα ε, περιέπλεκαν την ε, υπόθεση. Επίσης, άρθρο 4, εδώ η Κομισιόν προτείνει μια διάταξη για τους σκοπούς αυτής της πρότασης, Αναρωτιέμαι όμως, ο οργανισμός επισωτιών και τα σχετικά κριτήρια που υπάρχουν ε, δεν είναι καλύτερα γιατί είναι πιο πλήρη. Μετά, εδώ στο Κοινοβούλιο ε, έχουμε παράλληλες ε, διαδικασίες και δραστηριότητε και πρέπει και αυτό να το έχουμε υπόψη, να δούμε πώς θα Πώ θα κινηθούμε, να μην μιλούμε δηλαδή επί διαφορετικών νομικών πράξεων, να μην φτιάξουμε και κενό και να μην μπλέξουμε και σε, στη γραφειοκρατία. Γιατί μιλούμε και για την ε, εμπορική, για την πώληση των ε, ζώων συντροφιά, ε, Υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο για την υγεία των ζώων και θα πρέπει εδώ να έχουμε σαφή όρια. Και επίσης πρέπει να είναι σαφές το τι ακριβώς θέλουμε να ρυθμίσουμε και τι θα κάνουμε με τα αντιβιωτικά. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, το οποίο βεβαίως ε, θα πρέπει να συζητηθεί στην έκθεση, αλλά βεβαίως είναι και πολύ ευρύ ως κεφάλαιο. Ε, επίσης έχουμε την αναθεώρηση των, ε, του κανονισμού για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Είναι σωστό αυτό, μήπως είναι λάθος, να το συζητήσουμε. Και το ίδιο ισχύει και κάποια άλλα σημεία. Έχουμε λοιπόν πολλή δουλειά, και, αλλά αν παραμείνουμε στην γραμμή που προτείνει η κυρία Πόλσεν, νομίζω ότι στο τέλος θα μπορούμε να είμαστε πολύ περήφανοι ως Κοινοβούλιο, γιατί θα έχουμε υποβάλει μια πολύ καλή έκθεση, η οποία είναι πάρα πολύ απαραίτητη και που τη ζητούμε εδώ και πολύ καιρό. Ευχαριστούμε και συγχαρητήρια κυρία Πόλσεν. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γέγκλε. Η κυρία Αγιούσο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια για την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Το πρώτο που θέλω να σας πω είναι να ευχαριστήσω την κυρία Πούλσεν για τις εξηγήσει της και θα πρέπει να, να πω ότι όντως εδώ πέρα δεν πρόκειται για ένα κανονισμό που αφορά την κατατοχή των ζώων και άρα εδώ πέρα θα πρέπει να προσέξουμε τι θέλουμε να τροπολογήσουμε. Η Επιτροπή προτείνει για το πώς θα βελτιωθούν οι σχετικές διατάξεις, πώς θα υπάρχει καλύτερος έλεγχος, εισαγωγή και κάποια άλλα ζώα. Και όπως και ο άλλος κανονισμός που αφορούσε τα φυτά και εδώ έχουμε είπαμε κατάχρηση των δυνατοτήτων για έκδοση ε, κατά εξοδότηση πράξεων στόχος όμως είναι σωστός, η βάση είναι σωστή και επομένω επιδέχεται βελτίωση το κείμενο. Και να δούμε τι θα γίνει με τις εκτελεστικές και τις κατεξιώδει πράξεις. Θα ήθελα όμως να μας ξεκαθαριστούν κάποιοι ορισμοί. Πρέπει να ξεκαθαριστεί τι είναι η ε, ζώο ε, ελεύθερο, τι είναι ζώο μη ελεύθερο, τι θα πει έλεγχος, άλλο ένα ζώο ελεύθερο και άλλο ένα ζώο σε εκτατική εκμετάλλευση την ιατρική. Τι είναι, είναι κάποιο σε άγρια κατάσταση. Με τον κόσμο αυτό επίσης θέλουμε να ελέγξουμε και τις επιζωοτίες αυτές που αφορούν ή έχουν πηγή τα άγρια ζώα. Κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα όσον αφορά τις εξαγωγές θα πρέπει να δούμε τι ισχύει από πλευρά ε, κτηνιατρική στα κράτη-μέλη ω προ τι τρίτε χώρε. Θα σα πω αυτό το οποίο είχα πει και για τα φυτά. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με τι αγωγέ ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε επίπεδο εθνικό το τι κάνει κάθε χώρα με τι τρίτες χώρε, Σε εξαγωγέ δηλαδή τη κάθε χώρα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηριχθεί με την κοινή προσπάθεια αυτή που θα κάνει το άρθρο 9, θα πρέπει να το ξαναδούμε, που λέει για όλους τους αλωσομένους, λέει για αυτούς που θα πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν γνώσεις στον δομή της υγείας των ζώων. Θα πρέπει να το χτενίσουμε το σχετικό άρθρο. Εδώ καλύπτω και τα άγρια ζώα, πάρα πολύ δύσκολο να τα ελέγξουμε βέβαια. Αδύνατον ουσιαστικά να τα ελέγξουμε. Δεν δυνατόν να υπάρξουν κανόνες για να τα υποπτεύουμε. Τώρα όσον αφορά την επισήμανση κινδύνων προτείνεται ε, να δούμε πώς θα ρυθμίσουμε τις πληροφορίες πιστεύω και όχι την μορφή των πληροφοριών γιατί κάθε χώρα έχει δική της μορφή πληροφοριών και ενημέρωση. Όταν κανείς διαβάζει αυτή την πρότασή σας, η εντύπωση είναι ότι εσείς θέλετε να ελέγξουμε τις κινήσεις των ζώων σε κάθε κράτος μέλος. Ίσως και όχι, αλλά όμως εκ πρώτη όψεως θα πρέπει αυτό να είναι εθνική απόφαση, να το αφήσουμε αυτό μόνο στην επικουρικότητα. Dziękuję Pani Poseł. W tej chwili proszę o zabranie głosu το Chairman, the subject of this agenda... Το θέμα αυτού του σημείου της ημέρας της διάταξης είναι η, ε, ζωή των, υγεία των ζώων. Θεωρεί κάποιο ότι ε, ένα υγιέ ζώο ε, μάλλον θα παραμείνει και ζωντανό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία μάλλον, λέει ότι θα, μάλλον αν εισαχθεί στην, Ευρωπαϊκή, στην ε, Βρετανία θα σκοτώσει ε, εκατομμύρια πουλερικών κάθε χρόνο. Και αυτό προφανώς δεν είναι καλό, γιατί μιλώ για την αναβληθήσα απαγόρευση του εκοψίματος του ράμπου των πουλιών, των κοτόπουλων. Εγώ λέω ότι δεν είναι κάτι απλό αυτό. Δεν είναι απλώς ότι θα νιώσει κάτι, θα νιώσει μια μικρή έτσι, δυσφορία το κοτόπουλο, είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό. Με τις, γιατί αυτό γίνεται με υπέρυθρες ακτίνες. μπορεί να υπάρξει αιμορραγία και αν υπάρξει αιμορραγία πρέπει να ληφθεί όλο και περισσότερο ε, αίμα και στο τέλος καταλήγει κανείς να κανιβαλίζει το κοτόπουλο. Αυτό, σε αυτό καταλήγει. Εμείς προσπαθούμε στον Εμένο Βασίλειο να αποτρέψουμε αυτή την τρέλα, την ε, καλών προθέσεων τρέλα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιοι ε, παραγωγοί έχουν θελοντικά προσφερθεί να διατηρήσουν τα ε, σμήνη χωρίς να, τα, να κόψουν τα, ε, ε, ράμφη για, τις 14, για τους 14 μήνες που τα κρατούμε. Ε, αλλά τελικά τα παράτησαν και κάλεσαν κάποιους να ε, κόψουν τα ράμφη των πουλιών. Θέλουμε να αποφύγουμε λοιπόν τέτοια περιστατικά και θέλω η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει ε, να ασχολείται με το θέμα αυτό γιατί θα πάρει πολλά χρόνια να, για να μπορέσουμε να ε, μεγαλώσουμε νέα πουλιά που δεν θα είναι επιθετικά επειδή ακριβώ ε, τους, τα υποβάλλουμε σε τέτοιε διαδικασίες. Ας αφήσουμε λοιπόν την νομοθεσία που θα σκοτώνει ζώα. Ας δούμε μια νομοθεσία που θα βοηθάει τα ζώα. Ας βάλουμε λοιπόν κάπου ένα φρένο. Έχουμε εξαντλήσει λοιπόν τον κατάλογο των ομιλητών, λέει ο Πρόεδρος. Θα ήθελα να ζητήσω από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Αλμπέρτο Λαντομάδα, να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την εισηγήτρια και όλους εκείνους που πήραν το λόγο. Θεωρώ ότι ουσιαστικά εχαιρέτησαν ε, την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολύ φιλόδοξη είναι η πρόταση. Να επενθυμίσω ότι η πρόταση αυτή καταργεί και αντικαθιστά 40 νομοθετικά κείμενα του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου που υπάρχουν. Είναι ένα εγχείρημα νομικό περιπλοκότατο. Χρειάστηκαν πολλά χρόνια εργασία Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να ετοιμάσει την πρόταση. Σίγουρα η συνεισφορά του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα είναι σημαντική για τη βελτίωση της προτάσεως περαιτέρω. Μία από τις μεγάλες ανησυχίες, αλλά πρέπει να πω την περιμέναμε, είναι αυτή που αφορά το μεγάλο αριθμό κατεξοδότηση πράξεων και εφαρμοστικών πράξεων που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εδώ στρέφομαι σε αυτό που ήδη είπατε. Αυτή η πρόταση αντικαθιστά 40 νομοθετικά κείμενα τα 40 αυτά κείμενα έχουμε πολλές εκατοντάδες αναθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υιοθετεί δευτερογενή νομοθεσία. Σύμφωνα με το παλιό καθεστώς επιτροπολογίας. Από πολλές εκατοντάδες ε, πράξεις τις μειώνουμε στις 100-150 ε, συνολικά, όπως είπε και κάποιος ομιλητής. Γι' αυτό λέω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να είναι αναλογική στην προσέγγιση της. Όσον αφορά, πώς να το πω, την υποδιέρεση που προβλέπεται από τη συνθήκη της Εισαβόνα σε βασικές πράξεις, κατεξοδότηση πράξεις και εφαρμοστικές. Είμαστε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε και με το Συμβούλιο και, την Ευρωπαϊκή, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ακούσουμε το input τους Ακούσαμε ένα input όσον αφορά τον κατάλογο των ασθενειών. Με τα χαράς να συζητήσουμε μαζί το θέμα, πώς μπορεί να βελτιωθεί ο κατάλογος. Κάποια προβλήματα θεμελιώδη. Αυτή η πρόταση δεν αφορά την ευζοία των ζώων. Τη λαμβάνει υπόψη, όπως ζητήθηκε από τη συνθήκη, από το άρθρο 13, και υπάρχουν πολλές παραπομπές στην ευζοία των ζώων σε όλο το κείμενο. Όπου χρειάζεται κάτι τέτοιο, ξεκινώντας από κριτήρια. Η καλή μεταχείριση, η καλή αντιμετώπιση των ζώων είναι κάτι πολύ σημαντικό. αν έχει κάποια αρρώστια και έχει πληστεί η γλώσσα του μοσχαριού και το εμποδίζει να φάει και να μυρικάσει, υποφέρει. Άρα η έλλειψη ε, ασθενειών έχει σημαντική ε, επιρροή στην καλή διαβίωση του ζώου. Και αυτό το λαμβάνουμε υπόψη όταν θέλουμε να θέσουμε προτεραιότητες και να δημιουργήσουμε κατηγορίες όσον αφορά την παρέμβαση Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσον αφορά τον έλεγχο των σημαντικών ασθενειών. Άλλη πτυχή που αναφέρθηκε, που είναι πολύ σημαντικό, η αντίσταση στα αντιβιωτικά. Όσον αφορά το θέμα, ήδη υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο στην οδηγία, παραδείγματο χάρη, που ισχύει και τον κανονισμό για τον έλεγχο των ζωονόσων. Έχουμε δύο νομοθετικές πράξεις του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου που δεν, αντικαθιστούν, που δεν αντικαθίστανται από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθμίσεις, αλλά θέλουμε να εντάξουμε καλύτερα με την πρότασή μας την παρούσα προσέγγιση όσον αφορά το πρόβλημα της αντίστασης στα αντιβιωτικά. Αποσαφηνίζουμε όμως ότι οι δράσεις πρόληψης ελέγχου των παθογόνων φορέων που ανθίστανται στα αντιβιωτικά, αυτοί μπορούν να ελεγχθούν και ανεξάρτητα από την επίδραση που έχουν στην ανθρώπινη υγεία. Με άλλα λόγια, αν υπάρχουν φορείς νοσογόνοι που έχουν χαρακτηριστικά αντίσταση στα αντιβιωτικά, μπορούν να ελεγχθούν, πρέπει να ελεγχθούν ακόμα και αν αυτοί οι νοσογόνοι φορείς δεν πλήττουν τους ανθρώπους, αλλά φορούν μόνο τα ζώα. Άρα συμπληρώνουμε το νομοθετικό πλαίσιο. Βέβαια κάποιες πτυχές παραμένουν εξίσου εκτός του πεδίου εφαρμογή της πρότασής μας. Η σωστή χρήση των φαρμάκων είναι κάτι που ρυθμίζεται από από την νομοθεσία για τα φάρμακα. Δεν ρυθμίζεται από την νομοθεσία για την υγεία των ζώων, ούτε από την νομοθεσία για τον έλεγχο των μεταδοτικών ασθενειών, μεταδοτικών ε, ασθενειών των ζώων που μπορούν να μεταδοθούν στους ανθρώπους. Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία με τους συναδέλφους για την νομοθεσία για τα φάρμακα, ούτως ώστε να λαμβάνονται παντού όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προλαμβάνονται και να ελέγχονται στο βαθμό του δυνατού τα προβλήματα αυτά της αντίστασης στα α, αντιβιωτικά. Ένα πρόβλημα που αναφέρθηκε αφορά το εμπόριο. Πώς αυτή η πρόταση θα ρυθμίζει το εμπόριο. Ακούστηκε σχετικό σχόλιο. Αφορούσε σε εθνικό επίπεδο τη μετακίνηση των ζώων. Δεν αλλάζει η πρόταση την ισχύουσα κατάσταση. Βέβαια υπάρχει ρύθμιση ακριβέστατη σχετικά με την μετακίνηση και το εμπόριο ζώων μεταξύ κρατών μελών. Αφήνουμε όμως στη διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών τη ρύθμιση της μετακίνησης των ζώων εντός των συνόρων τους. Δεν αλλάζουμε λοιπόν την προσέγγιση. Όσον αφορά το πρόβλημα των εισαγωγών, το πρόβλημα αυτό ρυθμίζεται άριστα από την ισχύουσα νομοθεσία. Θέλουμε απλώς να ενισχύσουμε τις διατάξεις για την υγεία των ζώων, τις σχετικές με την εισαγωγή ζώντων ζώων, προϊόντων ζωικής προελεύσεως, Όσον αφορά τις εξαγωγές, αυτό που προτείνεται είναι η βελτίωση όχι μόνο η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά την υγεία των ζώων και η νομοθεσία αφορά την υγεία των ζώων, αλλά να βελτιωθεί και η κατανόηση από πλευρά τρίτων χωρών της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε επίγνωση του πόσο δύσκολο είναι να εξηγήσουμε σε τρίτες χώρες τη μοναδικότητα της Ένωσης, την περιπλοκότητα της νομοθεσίας μας. Αυτοί οι δύο παράγοντες, μοναδικότητα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και περιπλοκότητα της νομοθεσίας της, συχνά χρησιμοποιούνται από τρίτες χώρες ως δικαιολογητικά δικαιολογίες για να μην δεχθούν τα προϊόντα μας. Γι' αυτό θέλουμε από τη μία πλευρά να ενισχύσουμε τη θέση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, το στάτους της και από την άλλη να απλουστεύσουμε την νομοθεσία μας ούτως ώστε να γίνει πιο ευλήπτη από τις τρίτες χώρες. Τι ο τρόπος θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τις εξαγωγές μας. Κάποια απάντηση συγκεκριμένη τους ε, ομιλητές που παρενέβησαν. Τα εργαστήρια αναφοράς. Τα εργαστήρια αναφοράς που είναι 14 σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή και ασχολούνται με τις ζωονόσους είναι θεμελιώδη στοιχείο που βοήθησε πάρα πολύ την πολιτική για την υγεία των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη βελτίωση αυτής με την πάροδο των δεκαετιών. Τα εργαστήρια αυτά έκαναν δουλειά θεμελιώδου σημασίας για το συντονισμό των εθνικών εργαστηρίων. Και πώς να το πω, και να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη. Ήταν θεμελιώδη εργαστήρια ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην επιστήμη που είναι πίσω από την νομοθεσία για την υγεία των ζώων. Γνωρίζουμε ότι η πρότασή μας ενισχύει το σύστημα των εργαστηρίων αναφορά, συγγνώμη. Είναι παράλληλη πρόταση που υπάρχει, που είναι παράλληλη με τον προπολογισμό, που εκεί επιβεβαιώνεται τη Βούλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ένωσης στον προπολογισμό να ισχυροποιηθεί το σύστημα των εργαστηρίων αναφοράς. Υπάρχει και άλλη πτυχή που σχετίζεται με τα εργαστήρια όταν γίνεται λόγος στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πρώτη φορά στις τράπεζες διαγνωστικών αντιδραστικών φορέων. Το είδαμε σε κάποιες ασθένειες. Υπάρχει ε, δυσκολία να εντοπιστεί στην αγορά άμεσα μια λύση διαγνωστικών ουσιών που είναι θεμελιώδου σημασία για τη διάγνωση ασθενείας και συνεπώς για την πρόληψη και τον έλεγχο. Η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει τη δυνατότητα να δημιουργηθούν τράπεζε φορέων διαγνωστικών, ουσιών διαγνωστικών, που θα είναι τράπεζε που θα τις χειρίζονται τα εργαστήρια αναφορά, ούτω ώστε αυτά τα διαγνωστικά στοιχεία να τίθεται στη διάθεση των κρατών μελών, των εργαστηρίων των κρατών μελών σε περίπτωση ανάγκης. Οπότε σας επιβεβαιώνω ότι θέλουμε να ενισχύσουμε το σύστημα αυτό των εργαστηρίων αναφοράς. Όσον αφορά την ομοθεσία που αναφέρθηκε για τη σπογκώδη εγκεφαλοπάθεια, τις διάφορες ζωονόσους και τα υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης. Καλύπτει μέσω των βασικών αρχών η πρόταση και αυτή την νομοθεσία. Όμως όπως προανέφερα, σε σχέση με την αντίσταση στα αντιβιωτικά, δεν αντικαθιστά συγκεκριμένες ειδικέ νομοθετικές πράξεις, όπως είναι ο κανονισμός για τη σπογκώδη εγκεφαλοπάθεια, η οδηγία για τις ζωνόσους και ο κανονισμός για τα υποπροϊόντα, δεν αντικαθίστανται, ισχύουν όσον αφορά τη δημόσια υγεία. Και η δημόσια υγεία ε, είναι ανώτερη από την υγεία των ζώων. Δεν θέλαμε να έχουμε υπερβολικέ ε, φιλοδοξίε που θα ήταν επιζήμιε για την νομοθεσία. Οπότε προσπαθήσαμε όλα αυτά να τα καλύψουμε κατάλληλα. Δίνουμε σημασία στην κατάρτιση βέβαια. Θέλουμε να έχουμε παραγωγικό τομέα, κτηνιατρικό τομέα που να ασχολείται με επίσημους ελέγχους και άλλες επίσημες δραστηριότητες που έχουν ανατεθεί στον τομέα και να γίνονται όλοι πιο ικανές οι αρχές, οι αρμόδιοι φορείς. Δεν θα επισέδω σε λεπτομέρειες τώρα για κάποια άδεια ή κάτι άλλο. Αυτό είναι θέμα των διαφόρων κατοξισοδότηση πράξεων. Όποτε χρειάζεται αυτό. Όποτε χρειάζεται να κινηθούμε προς τα εκεί. Έλεγχος των ασθενειών στα άγρια ζώα. Δεν προτείνει η Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προτείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ενδιαφερθεί για όλες τις ασθένειες των αγρίων ζώων, αλλά υπάρχουν ασθένειες που προφανώς μπορούν εύκολα να μεταδοθούν από τα άγρια ζώα και εκτός των συνόρων των κρατών μελών και μέσω συνόρων των κρατών μελών με τίτες χώρες να μεταδοθούν. Έχουμε παράδειγμα με την πανόλη των χείρων από την Αφρική που μπορεί να διαδοθεί από Ρωσία και Λευκορωσία ε, μέσω των ε, αγριογούρουνων. Έχουμε κάποιες εμπειρίες όσον αφορά τον έλεγχο των ασθενειών των αγριών ζώων και θετικές εμπειρίες όπως ο έλεγχος της λύσας ε, στα όρνια μες, συγγνώμη, στις αλεπούδες. Λοιπόν, Θέλουμε λοιπόν να έχουμε καλό έλεγχο των ασθενειών των αγρίων ε, ζώων, χωρίς όμως να κάνουμε το αμάρτημα να είμαστε ε, πάρα πολύ ε, φιλόδοξοι. Πρόεδρε, εδώ κλείνω. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στη διάθεση της εισηγήτριας και οποιοδήποτε άλλου θέλει να εκφράσει την άποψή του για να συνεργαστούμε ε, και να φτάσουμε πιο γρήγορα στην έγκριση αυτού του κειμένου. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γέγκλερ θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα ερώτημα στην Κομισιόν μπορώ να θέσω. Η Κομισιόν έχει σκεφτεί πιο συγκεκριμένα για το ναι. σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τι θέλει να ρυθμίσει ακριβώς. Έχει συγκεκριμένα τμήματα μέσα σε αυτό το πακέτο τα οποία εμπίπτουν στην επικουρικότητα και άρα παραμένουν στη διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κανέναν άλλον να ζητάει το λόγο, οπότε να δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν για να απαντήσει. Thank you, Mr. Chairman. Ε, ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπε ο ε, πρόκειται εν πολλής εδώ για μία νομοθεσία που θέλει να καλύψει το πρόβλημα των μεταδοτικών ασθενειών. Γιατί, διότι αυτό το συμβαίνει εδώ, η υποκτήμενη αξία, είναι προφανής. Είναι αυτέ οι ασθένειε οι οποίε όντως είναι τα μεταδίδονται ε, μέσω των συνόρων και οπότε θα πρέπει αντίστοιχα να είναι εναρμονισμένη η αντιμετώπιση του, η καταπολέμησή του. Οπότε φυσικά αυτό το οποίο κάναμε ήταν να μπορέσουμε να επεκταθούμε, να διευρύνουμε τα κριτήρια όσον αφορά αυτέ τι ασθένειε. και ε, αυτό τώρα, τώρα σας το λέω εν συνόψη, να είναι σαφές για ποιες ασθένειες ε, γίνεται, ε, ε, επιβάλλεται κοινοτική δράση. Παρ' όλα αυτά, τα κράτη-μέλη θα έχουν περιθώριο μόνο τόσο ώστε να μπορέσουν να αναλαμβάνουν δράση ώστε να βρουν κάποιε άλλε ασθένειε. Υπό τον όρο βέβαια ότι ε, το τι κάνουν τα κράτη-μέλη δεν θα αντιβαίνει στι αρχέ του νομοθετήματο και δεν θα αντιβαίνει στι αρχέ τη ενία αγορά. Να μην ξεχνούμε ότι επί πολλέ δεκαετίε οι επιζωτίε είναι πρόφαση προσαρτησμού. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Και πάρα πολλές φορές οι τέτοιες χώρες προσπαθούν να περιορίσουν τις εισαγωγές τους επί τη βάση του ότι δεν υπάρχει επαρκή αιτιολόγηση, άρα θα πρέπει κανεί να είναι πάρα πολύ προσεκτικός όσον αφορά την ισορροπία μεταξύ του, της διαχωριστής του πού μπορεί να πανεβαίνει η Ένωση και πού τα κρατημέλη. Τα κρατημέλη επομένως θα πρέπει να διέπονται από κάποιους περιορισμούς, αλλιώς μπορεί να ολιστήσουμε στην κατάσταση αυτή της, ε, της χρησιμοποίησης τέτοιων δικαιολογιών για τον προστατευτισμό. Κύριε Γέγκλε. Από ό,τι βλέπω ανέβετε ε, με τρόπο δείχνει ότι είστε ικανοποιημένοι, ότι καλυφθήκατε. Τι Πόλσεν, αν θέλει μπορεί να λέτε το λόγο. Ναι, πρόεδρε, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ πολύ τους ε, συναδέλφους και ιδίω τους σκιώδους που το λόγο. Νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς να συνοψίσει τα συζητηθέντα. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι ακόμη σαφέστερα από ό,τι προηγουμένω. Ναι. Ότι θα πρέπει να κινηθούμε σε αυτό το πλαίσιο. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις μεταδικές ασθένειες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι έτσι θα κάνουμε σημαντικά βήματα πρόοδου και επίσης θα συνεργαστούμε πάρα πολύ καλά με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Επίσης, θα ήθελα κάτι άλλο να προσθέσω στον αφορά του Σκιώδη, συζητάς. Για τις επόμενες 15 μέρες πρόκειται να απουσιάζω. Θα σας πω άλλη φορά. Πού θα πάω, γιατί θα κάνω από αρχάς Οκτωβρίου, πότε να αρχίσει στην πραγματικότητα η δουλειά μας. Ελπίζω να πάμε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Εισηγήτρια. Θα έχουμε μία ακρόαση για το θέμα αυτό στις 25 ε, Νοεμβρίου. Και επίσης άλλο ένα, άλλη μια τέτοια ακρόαση στις 5 Νοεμβρίου. Κυρίε και κύριοι, καλύψαμε τη σημερινή ημερησία διάταξη. Μια που γνωμοδότηση του κυρίου Σιλβέστρη δεν θα ζητηθεί σήμερα, βλέπει η ζήτησή τη. Οπότε έχω κάποιε ενδιαφέρουσε πληροφορίε. Η Κόπα Κοζεκά θα σας ε, καλέσει σε ένα κοκτέιλ. Απόψε. στις 6 ώρες εδώ στο Κοινοβούλιο. Εδώ στην αίθουσα, εδώ στην αίθουσα ε, 3G. 6 ώρα, όχι νωρίτερα. Πρόσκληση επαναλαμβάνω της Κόπα Κοζεκά. Εδώ, εδώ, μπροστά στην αίθουσα που βρισκόμαστε. Μάλλον εδώ στο 5G3, στην αίθουσα που βρισκόμαστε, εδώ απ' έξω, εκεί είστε καλεσμένοι. Έχει αρχίσει αυτή η εκστρατεία, ξέρετε, που ονομάζεται η σημασία της γεωργιας Τέτοια μερικη εκστρατεία που έχει μέσω του Ιντερνετ, μέσω των ε, μέτρων κοινωνική δικτύωσης, ε, στο μετρό, παντού. Εκεί λέει για τους αγροτικούς εταιρισμούς πόσο σημαντική είναι για την ε, της αγροτικής πολιτικής, για την διατροφική ασφάλεια. Οπότε και σήμερα για αυτό το λόγο θα γίνει αυτό το κοκτέιλ γιατί ολοκληρώνεται αυτή η πανημερωτική εκστρατεία. Επίσης θα απονομηθούν και κάποιοι έπαινοι κάποιο είδου βραβεία. Θα μας μιλήσει ο κ. Δεκάστρο για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθη επί της ΚΑΠ. Θα μιλήσουμε για την γενικότερη σημερινή κατάσταση και επαναλαμβάνω ότι και ο επικεφαλής της ΚΟΠΑΚΟΖΕΚΑ θα ε, μιλήσει, ας πει τη γνώμη του για το τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Γεωργία, σήμερα στο κοκτέιλ που έχουμε προκεκλημένοι εδώ έξω από αυτήν εδώ την αίθουσα. Στις 6 ε, ώρα. Είστε προσκεκλημένοι. Σας προσκαλώ έξω τη Κόπα Κοζεκά. Ε, δεν περιμέναμε να τελειώσουμε τόσο νωρίς, αλλά τι έγινε. Έτσι, τελειώσαμε την ημερησία διάταξη. Έχετε κάτι να ρωτήσετε, κάτι να σχολιάσετε. Οπότε κύριε το πέρα της συνεδριάσεως και θα τα πούμε αύριο εις τις 9. Και θα σε ενημερώσω για τις αλλαγές στη μέση διάταξη. I είδες όλες all is clear. I think that's all is clear. Yeah, yeah, yeah.